Καλημέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχετε το μέγα πλεονέκτημα και προνόμιο να προεδρεύει η πρεσβυτέρα εδώ των βουλευτών, διότι έχουν όλοι ανηλυμένες υποχρεώσεις, κυρίως η πρόεδρος μας που πρέπει να ασχοληθεί με το πακέτο για τη διακυβέρνηση, τη δέσμη των 6 μέτρων, αυτό το six pack που δεν είναι καφάση μπύρε, αλλά είναι άλλο πράγμα. Έγκριση ημερήσια διάταξη. Έχει κανεί τίποτα να πει για την ημερήσια διάταξη. Όχι, εγκρίνεται. Δεύτερον, ανακοινώσει πρόεδρου εγώ δεν έχω. Ούτε εκείνη έχει, αφού απουσιάζει. Πάμε μέσα στην ακρόαση τώρα. για τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Καλωσορίζω στη δημόσια αυτή ακρόαση για το ΣΕΠΑ, για τα εμβάσματα και τις άμεσες ε, εκταμιεύσεις. Ξέρετε ότι είναι η πρώτη φάση Κάποιοι θα θεωρούν ότι είναι η εισαγωγή του ευρώ σε πληρωμές ε, διαφορετικές από μετρητά. Δύο ψηφίσματα έχει κάνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 και το 2010 που καλούσαν για αποφασιστικά βήματα προς την επίλυση αυτού του θέματος. Καλωσορίζω λοιπόν τους ομιλητές μας, την κυρία Γκέτρουτ Τούμπελ Γκούγκερελ, είναι μέλος του ε, Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έκλεισε το μικρόφωνο τη Πρόεδρου. Uh, uh, uh, Δυστυχώ δεν θα μπορέσει να παραμείνει μέχρι το τέλος της ακρόασης η κυρία Τούμπελ Κούγκερελ και θα παρακαλούσα να κάνετε τις ερωτήσεις σας αμέσως μετά την παρουσίασή της στη σύντομη συζήτηση που θα ακολουθήσει και γνωρίζετε ότι η ακρόση αυτή θα είναι η τελευταία επίσκεψη της κυρίας Τούμπελ Γκουγκερέλ υπό την σημερινή της ιδιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εύχομαι, σας εύχομαι καλή σύνταξη Νομίζω ότι σας αντικαθιστά άνδρας, πράγμα που δεν μ' αρέσει. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είχε η ζωή. Και για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, θα σας δώσω μέσω στο λόγο. Για την τελευταία παρέμβαση στο Κοινοβούλιο. ποιόν μας, υπό την παρούσα ιδιότητα, ούτε κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έρχεται ξανά με άλλη ιδιότητα. Merci beaucoup, Madame Um, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου τιμή να σας μιλήσω και πάλι για το ΣΕΠΑ. Να σας θυμίσω το πλαίσιο. Πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι της ε, λιανικής ε, των λιανικών συναλλαγών του τραπεζικού συστήματος, 20 με 30% των συναλλαγών ε, δηλαδή, και αυτό που χρειάζεται είναι ένα ανταγωνιστικό επίπεδο υπηρεσιών και σταθερά μοντέλα επιχειρηματικά για τους παρόχους των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ακόμα ενιαία αγορά και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι υπηρεσίες πληρωμών θα υποστούν μια περαιτέρω μετα... Ε, ε, μεταρρύθμιση σε σύγκριση με τα όσα έγιναν τα περασμένα χρόνια. Θα δούμε περισσότερες καινοτομίες, μια, ε, μια μεγάλη ζήτηση για, για άνετες υπηρεσίες, αλλά και αυξανόμενες ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια. Αν μπορούσα να σας δώσω μόνο ένα μήνυμα απόψε, θα ήταν να κλείσουμε το φάκελο ΣΕΠΑ, ας εστιάσουμε την προσοχή μας στην καινοτομία, την επάρκεια και την ασφάλεια. Και αυτό που χρειάζεται για να κλείσει ο φάκελος ΣΕΠΑ ε, θα το σας το εξηγήσω σε λίγα λεπτά. Καταρχήν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες και την ισχυρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των ψηφισμάτων του πριν από δύο χρόνια, πριν από ένα χρόνο, αλλά και με τη δουλειά που έγινε του τελευταίο, τους τελευταίους μήνες στην προπαρασκευή μιας νομοδότησης που είναι πολύ σημαντική και θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Τι χρειάζεται. Χρειαζόμαστε διάφορα βήματα εναρμόνισης που έγιναν και στο παρελθόν Νομίζω πως ο κλάδος έχει εργαστεί όσον αφορά δηλαδή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα όσα επιτεύχθηκαν ε, πέντε σημεία. Έχουμε ένα φόρματ για τους αριθμούς ε, ε, λογαριασμών πληρωμών, έχουμε σύμμορφες υποδομές με το ΣΕΠΑ και έχουμε και ένα νομικό πλαίσιο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο μέσω της οδηγίας για τις ε, υπηρεσίες πληρωμών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικά, αλλά αν δούμε την ε, μετακίνηση προς το σύστημα ΣΕΠΑ είναι σχετικά μικρή. Ορισμένες ε, χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Σλοβενία αλλά και το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι ένα από τις χώρες που είναι πρωτοπόρες στην μετακίνηση προς το σύστημα ΣΕΠΑ και η Ισπανία βελτιώνεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχω δει και τα στοιχεία από τη Φιλανδία όπου υπάρχει μεγάλη πρόοδο. Αν δούμε όμως, ε, τα, ε, μάλλον αν δούμε τα κράτη που δεν είναι στην Ευρωζώνη θα δούμε πως το ΣΕΠΑ ε, ισχύει για 31 χώρε, δεν είναι μόνο για την Ευρωζώνη και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, τα εμβάσματα που γίνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, ήδη στο 82% τους ακολουθούν το φόρματ ΕΠΑ το ίδιο και για την ε, Δανία. Ε, είναι πολύ σημαντικό φυσικά, σπουδαίο αυτό φυσικά και νομίζω πως αυτές οι χώρες που έχουν προχωρήσει τόσο πολύ ωφελούνται από τις νέες αυτές υπηρεσίες και επίσης περίφωνος αριθμός IBAN ε, η μπαν ε, που συχνά συζητείται από τον κόσμο υπάρχουν χώρες όπου το IBAN είναι ένα, μια, ένα είδος ταυτότητας και στην Ιταλία χρησιμοποιείται τότε δηλαδή, ήδη. Δεν είναι και τέτοιο μεγάλο θαύμα να μετακινηθούμε προς αυτό το σύστημα. Τι είδαμε τα τελευταία χρόνια βέβαια, ε, ε, η αυτορύθμιση έχει τα ωριά της, όπως σας είπα ο κλάδος έχει κάνει πολλά, έχουν κάνει προτάσεις και προτείνει λύσεις, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια και νομίζω πως τώρα η νομοθεσία θεωρείται από όλους όσους αναμειγνύονται στην διαδικασία αυτή ως ε, μια απαραίτητη στήριξη για τη συμπλήρωση της μετάβασης στο σύστημα ΣΕΠΑ και τέλος ώστε να μικρύνει η περίοδος μεταφοράς σε αυτό το σύστημα. Πρόταση της Κομισιόν για τον κανονισμό πρόκειται για τεχνικές ε, προδιαγραφές που δεν είναι επίμαχες, οι διορίες για την μεταφορά σε αυτό το σύστημα. Ε, νομίζω ε, στηρίζεται η πρόταση για μια δωδεκάμινη, ε, ένα δωδεκάμινο χρονικό διάστημα για την μεταφορά στην ΣΕΠΑ, αλλά υπάρχει και η εναλλακτική της μιας μετάβασης μόνο. Είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να καταλάβει ότι χρειάζεται σαφήνεια σε αυτό το θέμα αυτό και ότι αν μείνει εκτός του κανονισμού δεν θα υπάρξει, δεν θα είναι σωστή λύση. Ένα επίμαχο θέμα είναι κατά πόσο η Κομισιόν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τον κανονισμό. Νομίζω πως εδώ εμείς υποστηρίζουμε την άποψη της Κομισιόν ότι το να έχουμε κάποια σε τεχνικές απαιτήσεις στο παράρτημα θα βοηθούσε ώστε οι τροποποιήσεις να γίνονται πιο εύκολες και αυτό το υποστηρίζουμε. Η χρέωση της, των συναλλαγών, το ήδη το ανέφερα. Δημοσιεύσαμε μια γνωμοδότηση πριν από μια εβδομάδα που αναφέρονται όλα τα στοιχεία. Υπάρχει ισχυρή στήριξη για την ολοκλήρωση του κανονισμού και υποστηρίζουμε και το περιεχόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η άμεση πίστοση. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ε, πρόοδος μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, γιατί αυτό θα προσέφερε πιο εύκολες υπηρεσίες, πιο άνετες υπηρεσίες για πολλές ευρωπαϊκές χώρες που δεν χρησιμοποιούσαν ένα, μια τέτοια γρήγορη υπηρεσία. Είναι επίσης και ασφαλές μέσο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσουμε το θέμα ώστε να υπάρχουν μεγαλύτεροι όγκοι σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών πληρωμών. Η μεταφορά στο σύστημα και τα στοιχεία εμείς υποστηρίζουμε την 31η Ιανουαρίου και για το, την χρέωση τα, την, ε, γιατί δεν, δεν χρέωση δεν υπάρχει ακόμα κάποιος ε, κανόνας και για την Κομισιόν πιστεύω πως θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να εμπλέκει τους διαμπλεκόμενους ε, φορείς, να υπάρχει σαφής διαδικασία για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ε, η συμμετοχή τους σε τα διάφορα βήματα. Για τις μεγάλες πληρωμές θα πρέπει να υποκλείονται από τον κανονισμό. Οι μεγάλες πληρωμές θα είναι επίσης σύμμορφες προς την ΕΣΕΠ, αλλά είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή. Για να ολοκληρώσουμε, η πρότασή μας είναι πολύ σημαντική ε, για αυτήν την ε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και την ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντικό για τις ε, υπηρεσίες πληρωμών αλλά και για να καταστεί η βιομηχανία πιο ανταγωνιστική και να εστιάσει σε πανευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί το θέμα μόλις αυτό θα είναι εφικτό και να δημιουργηθεί σαφήνεια όσον αφορά τις τελικές διορίες για αυτό το πρόγραμμα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Όπως σας είπα, έχετε την ευκαιρία να κάνετε τώρα μέσω ερωτήσεις την κυρία ε, που πρέπει να φύγει. Ή τώρα ή ποτέ λοιπόν. Κάντε τις ερωτήσεις σας. Αν έχετε τελειώσει θα φύγει. Δεν έχει ζητήσει ακόμα κανείς το λόγο. Η κυρία Ισαΐα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, δώσει εξουσιοδότηση για αποφάσεις σε κάποιους ενδιαφερομένους, αυτούς πώς θα τους συμβουλεύετε, θα πρέπει να είναι ένα συγκροτημένο σώμα, υπάρχει το Συμβούλιο ΣΕΠΑ, εκεί θα πρέπει να γίνεται κοστή η φωνή τους, είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους ακούμε κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Πού θα τους ακούμε αυτούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται πολύ να δίνει κατεξουσιοδότηση ε, πράξης. Θέλουμε εμείς να έχουμε την νομοθετική εξουσία στα χέρια μας. Πού νομίζετε λοιπόν θα γίνει αυτό, πού θα τους ακούμε και θα τους φερόμαστε εξίσου με το Κοινοβούλιο. Βεβαίω το Συμβούλιο ΣΕΠΑ που θεσπίστηκε πριν από ένα χρόνο θα ήταν το ιδανικό βήμα για να διοργανώνεται η συζήτηση ανάμεσα στον κλάδο, τι αρχές και του εκπροσώπους των καταναλωτών, επίσης ε, εκπροσώπους του δημόσιου τομέα. Νομίζω πως θα ήταν αυτός ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Πέρα από τη διαβούλευση, ε, τη δημόσια διαβούλευση, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα καλό βήμα. Äh, ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκλίντς. έχω μια ερώτηση για το δημόσιο τομέα. Είχα την εντύπωση ότι στη μεταφορά στο νέο σύστημα ο δημόσιος τομέας δεν ακολούθησε με τους ίδιους ταχύς ρυθμούς που θα περίμενε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που θα ήταν και προς το συμφέρον της μετάβασης στο σύστημα τι έγινε τώρα, βελτιώθηκε η κατάσταση ή διαφέρει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα ακόμα, παραμένουν οι διαφορές. Είναι διαφορετική η κατάσταση στις διάφορες χώρες αρκετά. Έχουμε δει πρόοδο σε κάποιες, ενώ σε κάποιες άλλες λιγότερο. Αν είναι πολύ καλά οργανωμένο το εθνικό επίπεδο, με φόρουμ ε, τοπικά ή περιφερειακά για τη ΣΕΠΑ, οι χώρες αυτές λοιπόν που έχουν προχωρήσει περισσότερο εποφελούνται σαφέστατα περισσότερο. 14% είναι η μεταφορά του δημοσίου τομέα στο σύστημα, αλλά το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες εργάζονται πολύ σκληρά για να ε, περάσουν και οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο σύστημα αυτό. Και έχει και συμπληρωματική ερώτηση ο κύριος Κλίντς. Μεγάλες επιχειρήσεις όπως ε, η ΕΝΤΕΦ Λιονές Δεζό μου στέλνουν λογαριασμούς ε, για το εξοχικό μου. Και του είπα τι μου στέλνετε για το ρεύμα, για το νερό λογαριασμό. Αν τα παίρνετε από το γερμανικό μου λογαριασμό απευθεία. Μου λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ψάξατε αυτό. Για ποιο λόγο δεν γίνεται. Γιατί εμεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πολύ γρήγορα ε, περάσαμε στο σύστημα ΣΕΠΑ και λειτουργεί πολύ καλά γιατί τα μέλη του προσωπικού μα ε, κατάγονται από διάφορε χώρε και μπορούν ήδη να χρησιμοποιούν του λογαριασμού στα κράτη του. Η κυρία Λούλινγκ χωρί μικρόφωνο. Oh, äh, Άλλες ερωτήσεις έχετε? Ναι. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τούρπελ και πάλι ό,τι επιθυμείτε για το προσεχές μέλλον και μπορεί να σας ξαναδούμε ποιος ξέρει το 2014-2019 θα τα δούμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Bon, on va continuer Συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα την κυρία Αν Φίλη. Αν Φίλη. που είναι επικεφαλής ε, του νομικού και οικονομικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης ε, Καταναλωτών και θα μας παρουσιάσει τη θέση των καταναλωτών και στη συνέχεια θα ακούσουμε και εκείνους που ε, αναπτύσσουν και προμηθεύουν τέτοια συστήματα πληρωμών, τον κύριο Γκέρχαρτ Χάρτσινγκ που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών και αντιπρόεδρος ε, στην ABN Άμρο για θέματα υποδομών και αγορών. Στη συνέχεια την κυρία Βαντχεφέρ που είναι πρόεδρος ε, της ομάδας εμπειρογνωμόνων και εργάζεται στη City Global Διευθύντρια και η κυρία Ναρίντα Βιγέ είναι επικεφαλής ε, των σχέσεων στρατηγικής και διατραπεζικών ε, των ε, κοσμίων γενικών συστημάτων πληρωμών στη Γαλλική Τράπεζα Κρεντή Αγρικόλ. Στη συνέχεια θα γίνει ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων και συζητήσεων με τα μέλη. Θα ήθελα και πάλι να θυμίσω σε όλους Ε, να ε, σέβεστε τους χρόνους σας ή δυνατόν να μην τους ξεπερνάτε. Δέκα λεπτά η κυρία Φιλή, οι υπόλοιποι τρεις, επτά λεπτά έκαστος. Ευχαριστώ. Και σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο σας. Η κυρία Φιλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να προειδοποιήσω τους διερμηνείς ότι άλλα έδωσα και άλλα θα πω. Ευχαριστώ την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ε, για την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Ενώσεων Καταναλωτών σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για τη ΣΕΠΑ θα εορτάσουμε την 50η επέτειό μας του χρόνου και εκπροσωπούμε στις Βρυξέλλες τις βασικές ενώσεις καταναλωτών ε, από 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η πρόθεση των ε, ενδιαφερόντων και συμφερόντων των καταναλωτών στις λιανικές πράξεις ε, τραπεζικές συναλλαγές μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ΣΕΠΑ η δημιουργία του χώρου, ενιαίου χώρου πληρωμών στην Ευρωζώνη, ε, ΣΕΠΑ, παρουσιάζεται εξίσου σημαντική όπως και η έλευση του ευρώ το 2002. Ε, τα εθνικά βάσματα τώρα θα μεταφραστούν σε πληρωμές παντού στην Ευρωζώνη. Ε, και υπάρχει μετάβαση λοιπόν προς αυτό το σύστημα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα καταρχήν για να δούμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο εύκολα ακόμα όπως θα θέλαμε. Βέλγιο, Γερμανία, ε, Γαλλία πρώτα. Η Μπεν Πεπαριπά, μεγάλη γαλλική τράπεζα και η πρώτη ε, βελγική ε, φόρτις έχουν συνενωθεί. Μπεν Πεπαριπά φόρτις. Εάν έχετε λογαριασμό σε βελγική τράπεζα 30 ε, λεπτά κοστίζει το έμβασμα. Ενώ 3 ευρώ και 40 στη Γαλλία. 11 φορές περισσότερο για μια βασική, ουσιαστική και αντίστοιχη τραπεζική πράξη de Πώς γίνεται αυτό μέσα στον ίδιο όμιλο να είναι τόσες οι διαφορές και πού είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΠΑ ή ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΠΑ αν ακόμα και στην ίδια τράπεζα ή στον ίδιο όμιλο διαφέρουν τόσο πολύ οι χρεώσεις. Ε, η ΣΕΠΑ επίσης ε, δεν ήταν ε, το βασικότερο που θέλουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές έτσι κι αλλιώς σε περισσότερες περιπτώσεις εθνικά εμβάσματα κάνουν. Η πρόεδρο, μήπω θα μπορούσατε να μιλήσετε λίγο πιο αργά γιατί δεν σα παρακολουθούν οι διερμηνείς ε, για λόγου ταχύτητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δύσκολο ε, να διαφημίσουμε τις ΕΠΑ ε, στα μάτια των καταναλωτών βασιζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Η υποστήριξη λοιπόν των καταναλωτών και των ενώσεών τους για τη ΣΕΠΑ ε, προέρχονται περισσότερο από μία πίστη τους στην ε, γενική ευρωπαϊκή οικοδόμηση και μια επιθυμία και ευχή επιτέλους να δουν μια ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών νικής. Ακόμα απόρο απέχουμε από αυτή την κατάσταση, αν το δούμε από τη σκοπιά των καταναλωτών. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε αν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μέσω πρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα έχουν πραγματικά πλέον εκτήματα από τη ΣΕΠΑ. Αν θέλουμε όμω να δώσουμε ευκαιρίε ε, στο σύστημα θα πρέπει να συντρέχουν διάφορε προποθέσει. Πρώτον, να ε, κυκλοφορούν ε, στην αγορά υπηρεσίε πληρωμών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκε και τα αιτήματα των καταναλωτών. Και επίση στη συνέχεια θα αναφερθώ σε αυτό να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε τον τρόπο λειτουργία και διακυβέρνηση τη ΕΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δούμε τι περιμένουν οι καταναλωτέ, Για να του πείσουμε να αλλάξουν από σήμερα ή πάρα πολύ σύντομα ε, τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα εθνικά του εμβάσματα και κατά τα άλλα είναι ικανοποιημένοι και να τα ανταλλάξουν με ε, πληρωμέ ΣΕΠΑ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Ευρωπαίο καταναλωτή να είναι πεπισμένο ότι αυτέ οι νέε υπηρεσίε πληρωμή ε, έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία εύλογα και θεμητά περιμένει. Και αυτά είναι τα τρία. Ε, τρία. Πρώτον, να είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, οι πληρωμέ να γίνονται χωρί λάθη και εγκαίρω. Δεύτερον, θα πρέπει αυτές οι υπηρεσίες πληρωμών να είναι ασφαλείς. Ε, είναι πολύ περιορισμένο το ε, ρίσκο της απάτης, αλλιώς ε, κινδυνεύει η αξιοπιστία. Γιατί τελικά την πληρώνει ο καταναλωτή, ο τελικό καταναλωτή και την απάτη. Και τρίτον, θα πρέπει να μην είναι ακριβέ αυτέ οι υπηρεσίε. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι ε, περισσότερε αυτέ οι υπηρεσίε πληρωμών οι καταναλωτέ τι θεωρούν βασικά προϊόντα. Καθημερινά κάνουν τι αγορέ του, πληρώνουν του λογαριασμού του. Δεν τα θεωρούν προϊόντα πολυτελείας για να έχουν υψηλά ε, ποσοστά κέρδου για τι τράπεζε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εμβάσματα και ε, τις αναλήψεις είναι ικανοποιητική η κατάσταση όχι μόνο λόγω του περιεχομένου του ε, κανονισμού αλλά και γιατί χάρη σε αυτό τον κανονισμό ε, γίνεται ε, ένα σύστημα γενικού ενδιαφέροντος στο ΣΕΠΑ και φεύγει από την περιορισμένη εφαρμογή που είχε στην αρχή. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Τα εξή τέσσερα σημεία είναι σημαντικά για μας. Πρώτον, δύο ε, διορίες για τη μετάβαση στο σύστημα. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την αρχή δύο καταληκτικές προθεσμίες. Ε, για τα εμβάσματα από το εθνικό στο ΣΕΠΑ γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, γιατί τα εμβάσματα περίπου είναι αντίστοιχα σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή αυτό το σύστημα ΣΕΠΑ μπήκε νωρίτερα στην αγορά, το γνωρίζουν περισσότερες, ε, περισσότεροι καταναλωτές. Αλλά για τις αναλήψεις τώρα, ε, είναι μεγάλη αλλαγή αυτή και χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνος προσαρμογής στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ε, άλλο θέμα. Υποστηρίζουμε όλα τα μέτρα που αποσκοπούν ε, στο να αποκτηθεί αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει αυτό ως προς την ασφάλεια των πληρωμών. Ένα τρίτο θέμα που χωράει η βελτίωση είναι όταν γίνονται αναλήψει με σταθερά ποσά δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, ε, αποζημίωση. Ο κανονισμός αυτός είναι μια ευκαιρία να αλλάξει το κείμενο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης να περιοριστεί η ε, μία αποζημίωση και να περιοριστούν επίσης καταχρήσεις συνέχεια. Ένα θέμα επίσης ενδιαφέρον ε, είναι οι ανταλλαγές. Βέβαια, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι ε, αμέσω ενδιαφέροντο ή προτεραιότητε για τι ενώσει καταναλωτών, αλλά οι ενώσει καταναλωτών είναι υπέρ διαφανών συστημάτων που θα επιτρέπουν στου καταναλωτέ να καταλαβαίνουν τι πληρώνουν και με άμεσο τρόπο και με έμεσο και ε, τι υπηρεσίε ε, παρέχονται. Το σημερινό σύστημα είναι διαφανές και παραπλανητικό εμπολής ε, για τους καταναλωτές γιατί καμιά φορά είναι πολύ ψηλές οι προμήθειες που παίρνουν οι τράπεζες ε, σε σχέση με το πραγματικό κόστος της συναλλαγής. Και αυτό που αγνοεί ο καταναλωτής είναι ότι το πληρώνει ο ίδιος τελικά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζει. Μόνο σε έξι κράτη-μέλη υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές πληρώνουν για τις αναλήψεις κάποιες προμήθειες που χρεώνουν οι τράπεζες. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτείνει ένα σύστημα προμηθειών σε περίπτωση απόρριψης, αντίρρησης επιστροφής της πληρωμής και ακύρωσης. Επίσης, δεν υπάρχει λόγος γιατί να πληρώνουν ε, τις επενδύσεις ΕΠΑ οι καταναλωτές και ακόμα περισσότερο αυτές τις αναλήψεις όταν δεν είναι οι ίδιοι ε, δικαιούχοι. Και ένα τελευταίο, πώς θα γίνει η διακυβέρνηση του ΣΕΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την τυποποίηση από την αρχή είναι πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη ισορροπίας, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών έχει ως μέλη του μόνο εκείνους που παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμών. Υπάρχει και το αντίστοιχο φόρουμ, αλλά αυτό είναι μόνο συμβουλευτικό όργανο και μόνο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών ε, είναι κυρίαρχη να παίρνει αποφάσεις. Εμείς έχουμε συμμετάσχει σε πολλές διαβουλεύσεις, σε πολλές συνεδριάσεις. Τελικά μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα επίλυσης διαφορών, διακανονισμού ε, ανεξάρτητο. Εμείς είχαμε να αποθέσει το Συμβούλιο ΣΕΠΑ κάποιες ελπίδες, αλλά αρνήθηκε να παίξει αυτό το ρόλο. Και θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως να είναι ευκαιρία αυτός ο κανονισμός για ένα οργανισμό ε, τυποποίησης ανεξάρτητο που να εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλα τα μέρη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αναλήψεις και για τις, τα εμβάσματα, γιατί ε, ε, διαγράφονται καινοτόμες ε, λύσεις και εκεί θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι φορείς από τις τράπεζες και μόνο. Τέλος, Πρέπει να σας πω ότι ανησυχούν για τις πληρωμές γενικότερα οι καταναλωτές, όχι μόνο για τη ΣΕΠΑ. Σας είπα προηγουμένως ποιες είναι ανησυχίες μας για τη ΣΕΠΑ. Ε, βράχει πρόθεσμα, βλέπουμε κάποιους κινδύνους τι γίνεται με τις κάρτες, ε, όχι τις πιστοτικές, τις χρεωστικές που, που είναι πολύ χρήσιμες και χρησιμοποιούν πολλοί καταναλωτές εντός ενός κράτους μέλους και μετά τι γίνεται με τον περιορισμό στην πρόσβαση σε μετρητά. Βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες είναι πολύ θερμή αυτή η συζήτηση. Έχουν γίνει κάποιες απόπειρες περιορισμού ε, της πρόσβασης ε, στα ATM. Πάντως, φαίνεται να αγνοούμε ότι πολλοί Ευρωπαίοι και πολλοί μετανάστες ε, δεν έχουν κάρτες, ε, μόνο μετρητά ε, χειρίζονται και σιγά σιγά αποκλείονται από την αγορά. Επίσης, τίθεται και ένα ζήτημα προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας του καταναλωτού, γιατί όταν κάποιος κάνει ανάληψη, κρατούν πολλά προσωπικά του στοιχεία. Αν θέλουμε οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν λιγότερα μετρητά, δεν θα πρέπει να τους δυσκολεύουμε την πρόσβαση στα μετρητά, αλλά να φθηνίνουν οι άλλες υπηρεσίες. Είναι πολύ νωρί ε, από τώρα να ε, προβούμε σε τέτοια μέτρα περιορισμού της πρόσβασης σε μετρητά. Τελειώνεται, λέει η Πρόεδρος. Ναι, η τελευταία φράση μου. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε μια επανάσταση στην υπηρεσία πληρωμών, αλλά όχι και επιταγή ελευκό. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά είμαι μόνη εκπρόσωπος των Χριστών εδώ σε αυτό το πάνελ. Ευχαριστώ. Συντόμευσα λίγο το κείμενο για να τηρήσω την προθοσμία των 7 λεπτών. Κυρίες και κύριοι, Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το διάλογο που έχουμε σήμερα. Όπως ξέρετε οι τράπεζες συνεργάζονται και έχουν συστήσει τα εναρμονισμένα συστήματα πληρωμών ΣΕΠΑ. Και βεβαίως ο στόχος δεν είναι να επιβάλλουμε στους πελάτες ε, το ΣΥΠΑ. Μάλιστα αυτό το απαγορεύει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τις κυβερνήσεις και τους ε, Ευρωπαίους ε, πολιτικούς. Οπότε καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαίου νομοθέτη να θέσει μια σαφή πρωτοβουλία για τη μετάβαση. Όμως έχουμε κάποιες ανησυχίες για την πρόταση κανονισμού της ε, Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μοντέλο άμεσης χρέωσης της ε, ΣΕΠΑ δείχνει πως ε, χρησιμοποιείται πάνω από το 75% των καταναλωτών που κάνουν σήμερα άμεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω από τα 17 δισεκατομμύρια άμεσων ε, πλήρωμων εμβασμάτων δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 γύρω στα 13 η 73% έγιναν στην Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσαν στην κοινή του επιστολή προ τα εμά στο ότι το ε, σύστημα ΣΥΠΑ βασίζεται σε αποδεδειγμένα εθνικά συστήματα, σέβεται πλήρω τι νομικέ απαιτήσει και ορισμένε φορέ πηγαίνει ακόμη και παραπέρα από αυτά τα οποία ορίζει η οδηγία περί πληρωμών. Τέλος. τρέπει ε, λοιπόν αυτό το σύστημα κάποια προαιρετικά χαρακτηριστικά που δίνουν την δυνατότητα να αντιδράσουμε στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Η πρόταση της Κομισιόν όμως σκοπεύει κάποια από αυτά τα προαιρετικά χαρακτηριστικά να τα κάνει υποχρεωτικά. Με άλλα λόγια η Κομισιόν θέλει να επιβάλλει σε όσους παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών να προσφέρουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούν το 75% των καταναλωτών και δεν τα ζητάνε. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν 4.000 τράπεζες που έχουν ήδη εφαρμόσει το σύστημα ΣΕΠΑ να επανεπενδύσουν στην ε, προσαρμογή των ε, συστημάτων τους. Άρα η τα εμβάσματα θα γίνουν άμεσα ή έμεσα πιο ακριβά για όλους τους ε, καταναλωτές. Και άρα αυτό αντιβαίνει το δεδηλωμένο στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πως η ΣΥΠΑ θα πρέπει να οδηγεί σε σταδιακή πτώση των τιμών. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Οδηγία οριστικοποιήθηκε μόλις πρόσφατα από τον Ευρωπαίο νομοθέτη για να υπάρχει ένα, ένα αρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του ΣΕΠΑ. Δεν υπάρχουν δείκτες για την ε, ανάπτυξή του. Το να γίνουν υποχρεωτικά χαρακτηριστικά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι προαιρετικά μπορεί να βλάψει τις ανάγκες των χρηστών γιατί μπορεί να θεωρήσουν πως είναι δύσχριστο το εργαλείο αυτό. Άρα η αγορά είτε θα πάει σε άλλα λιγότερα αποτελεσματικά συστήματα ή δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Η σωστή λοιπόν ισορροπία πρέπει να είναι αυτή μεταξύ της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Στο κοινή του επιστολή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν πως η αντιληπτή και η πραγματική ασφάλεια μπορεί να μην συμπίπτουν πάντα για να το καταστήσουμε σαφές. Το να γίνει υποχρεωτική αυτή η έλεγχη βασίζεται σε ένα σενάριο αντιληπτών κινδύνων που δεν ισχύει όσον αφορά την πραγματικότητα της αγοράς. Οπότε ο κανονισμός αυτός θα καταστήσει υποχρεωτικά αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή προαιρετικά. Δεύτερον, ανησυχούν πάρα πολύ όσον αφορά τις εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες που ζητάει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τροποποιεί μονομερώς ε, τεχνικές απαιτήσεις που υπάρχουν στο παράρτημα. Δεν χρειάζεται ούτε είναι αποτελεσματικό κανόνες των επιχειρήσεων και τεχνικές προδιαγραφές να ορίζονται διαρκώς και να επαναπροσδιορίζονται διαρκώς. Ούτε είναι δυνατόν η Κομισιόν να παίζει τον ρόλο ενός ε, project manager και να ορίζει προδιαγραφές. Όσον αφορά δε τις εκτελεστικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των τεχνικών απαιτήσεων μέσω πράξεων κατεξιοδότηση, δεν ε, καταφέρνει αυτή η πρόταση να εκπληρώσει ορισμένα βασικά κριτήρια, δηλαδή αυτό τη αναλογικότητας και της επικούρικότητα. Οπότε εμεί ζητάμε από τον νομοθέτη να αναγνωρίσει πως η αυτορύθμιση των τραπεζών στον τομέα των πληρωμών τα τελευταία 30 χρόνια σε γενικές γραμμές έχει αποδειχθεί ο πιο αποτελεσματικό τρόπο να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα εφικτό, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών. Θεωρούμε λοιπόν άρα πως τα άρθρα 12 έως 15 θα πρέπει να διαγραφούν από την πρόταση της Κομισιόν. Εάν όμω ο νομοθέτη αποφασίσει να δώσει αυτέ τι εκτελεστικέ εξουσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να διασφαλιστεί πως οποιασδήποτε απαιτήσει ε, τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τι συστάσει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού τη. Η δε πρόταση της ε, Κομισιόν για το ΣΕΠΑ περιλαμβάνει και τεχνικές προδιαγραφές και επιχειρηματικούς κανόνες που ισχύουν για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών. Βεβαίως, εμείς αναμειγνύουμε την, ε, εμείς, με καλωσορίζουμε την ε, πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρία να περιοριστούν μόνο στις τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, θα ήθελα να υπενηθήσω πως οι, υπηρεσίες πληρωμών είναι μια επιχειρηματική υπηρεσία, οπότε πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Επίσης το άρθρο 6 αναφέρει πως κανένα τέλος μυφ δεν η ανάλογη χρέωση δεν θα ισχύει για ε, τέτοιες ε, για τέτοια εμβάσματα. Οπότε εδώ πέρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της ε, θεμητής ε, εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να έχει ο ο επιχειρηματία ε, στην νομοθεσία. Η αρχή τη αναλογικότητα, όπω ορίζεται στο άρθρο 5 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει πω ε, η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ξεπερνά αυτό το οποίο είναι απολύτω απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι τη συνθήκη. Ο στόχος λοιπόν του κανονισμού ΣΕΠΑ είναι να περάσουμε από εθνικά σε πανευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών, κάτι δηλαδή το οποίο σημαίνει περισσότερο κόστος για τις εμπορικές τράπεζες και άρα δεν είναι απολύτως απαραίτητο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Θεωρούμε λοιπόν πως υπάρχει εδώ πέρα ένα λάθος στην κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την περιορισμένη ε, φύση του ανταγωνισμού για, την, ε, για τα πολυμερή τέλη που ισχύουν για τα εμβάσματα. Δεν εξηγεί η Κομισιόν πώς η ολοκληρωτική απαγόρευση τέτοιων ε, τελών μπορεί να ισχύσει επίσης και για πολυμερή και διμερή τέτοια τέλη για εθνικές συναλλαγές. Επίσης δεν εξηγεί γιατί αυτά τα τέλη διαφέρουν ουσιαστικά και δεν επιτρέπονται επί της αρχής σε αντίθεση με τα κανονικά πολυμερή τέλη συναλλαγών. Θεωρούμε λοιπόν πως δεν είναι προς το συμφέρον των ε, καταναλωτών να απαγορευτεί το τέλος αυτό το οποίο είναι maximum 8,8 Eurocents. Κλείνοντα, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω πως ε, έχει στηθεί το σκηνικό για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ΣΕΠΑ. Εμείς θεωρούμε πως αυτό ο στόχο θα πρέπει να παραμείνει το κέντρο της συζήτησης ε, στην αναθεώρηση του κανονισμού. Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο για τους ε, καταναλωτές, για όσου είναι παρόντες, στην είσοδο. Οπότε σας ευχαριστώ όλους που μας ακούσατε. Merci beaucoup. Euh, on passe tout de suite Ευχαριστώ πολύ. Ε, η Πρόεδρος θα δώσουμε αμέσως το λόγο στην κυρία Βαντχόφερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και την εισηγήτρια για την σπουδαία δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Να σας πω αμέσως γιατί είναι σημαντική η ΣΥΠΑ. Ένας ε, οικοδομικό, ένας οικοδομικός λίθος στο οικοδόμημα της ε, ενιαίας αγοράς. Μιλάμε για συναλλαγές 150 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω της ολοκλήρωσης αγοράς σε αυτό το επίπεδο, το ευρώ είναι ούτως ή άλλως μια πολύ σπουδαία φιλοδοξία από την έναρξη του ευρώ το 2000-2001 και υπάρχουν πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η πρόθεση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η πρόθεση της ψηφιακής ατζέντα και βέβαια η πράξη της ενιαίας αγοράς. Για τους χρήστες, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές, όπως ήδη είδαμε την παρέμβαση του κυρίου Κλίντς. Η ιδέα είναι να διευκολύνουμε ε, διασυνοριακέ άμεσε επιστώσει, ε, νέα υπηρεσία από την οποία θα πρέπει να ωφεληθούν και οι καταναλωτέ, και φυσικά για τι επιχειρήσει που λειτουργούν με ένα φόρματ και προδιαγραφέ κοινέ αυτό θα εξοικονομήσει ε, το, στο κόστο και θα βοηθήσει τι βιομηχανίε να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και θα προωθήσει το εμπόριο. Δηλαδή αυτό είναι και το όφελο του ενιαίου νομίσματος εξάλλου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε για να είναι επιτυχής αυτός ο κανονισμός. Θέλουμε να σας ε, υπογραμμίσουμε πέντε αρχές. Πρώτον, ε, η ενθάρρυνση της maximum εναρμόνισης. Θέλουμε πραγματικά να κινηθούμε από την εγχώρια ευρωζώνη, τα στάνταρ και τα φόρμα της σε πανευρωπαϊκές λύσεις, να υπάρξει ανταγωνισμός ανάμεσα στις τράπεζες και τους άλλους προμηθευτές πληρωμών, καθώς και τους ε, εκαθαριστές, τους οίκους μάλλον εγκαθάρισης ε, ενίσχυση της Ευρωζώνης, έπειτα ε, να μην υπάρχουν κόστη στις ε, συναλλαγές, ε, η υποχρέωση να εφαρμοστούν τα στάνταρ ISO σε όλη την η, μάλλον η επιβολή των στάνταρ ISO είναι ένα βήμα ε, περιττό κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη των πελατών μας. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε ένα ανταγωνιστικό ανοιχτό φόρουμ και συμφωνώ με την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την κυρία Σάια καθώς εκείνοι θεωρούν ότι το Συμβούλιο ΣΕΠΑ είναι το κατάλληλο βήμα για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων ε, φορέων και επίση ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο να προσαρμοστούμε αλλά να μην είναι και πολύ αργά ώστε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από την ολοκλήρωση σε μια ε, περίοδο μετά και την κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη βοήθησε στην επίλυση προβλημάτων. Πρώτον, ε, για την μέγιστη δυνατή εναρμόνιση, η πρόταση της Κομισιόν είναι κάπως δύσκολη όσον αφορά την άμεση αυτήν ε, ενέργεια ε, όσον αφορά την ε, εξοδότηση για τις τεχνικές προδιαγραφές σε αντίθεση με τις απαιτήσει της ΕΠΑ. Γι' αυτό και πρέπει να καθοριστούν όλα αυτά με ξεκάθαρο τρόπο οπότε δηλαδή θα πρέπει να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο εγχώρια όσο και διασυνοριακά. Διαλειτουργικότητα και προσβασιμότητα επίσης θα πρέπει να, να οριστούν καλύτερα ώστε να είναι σαφέστερες και θα πρέπει να υπάρξουν και Συγκεκριμένε προδιαγραφέ όσον αφορά τα εγχώρια προγράμματα και ποια από αυτά θα μπορούσαν να μπουν στο ΣΕΠΑ ή θα πρέπει να σταματήσουν μετά από μια κάποια μεταβατική περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει συμμόρφωση στο πλαίσιο το γενικό τη ΆΙΖΟ γιατί διαφορετικά τα φόρμα δεν θα είναι εναρμονισμένα και οι πελάτε δεν θα μπορούν να ωφεληθούν και να μπορούν να αλλάξουν εύκολα προμηθευτές δεδομένου ότι θα υπάρχει μια στάνταρ πρόσβαση τραπεζική. Η συγκήτρια ήδη έχει βελτιώσει το κείμενο σε πολλούς τομείς κλειδιά και εμείς προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μαζί της για αυτό το σημείο. Ανέφερα βέβαια το πεδίο εφαρμογή βασικά τα, μεγάλα συστήματα, τα, τα συστήματα μάλλον μεγάλων ε, πληρωμών καλύπτονταν από την νομοθεσία. Τώρα ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται, άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα το κόστος των συναλλαγών. Παρακαλώ αφού διαβάζετε, μην διαβάζετε τόσο γρήγορα. Οι καημένοι δερμηνείς δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Για το κόστος ε, με, της συναλλαγής είναι πολύ σημαντικό ε, της, μάλλον της μεταφοράς είναι σημαντικό οι πελάτες να μην χρειαστεί να πληρώσουν ε, το κόστος αυτής της μετάβασης και πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν είχε ε, διαβουλευτεί για την ε, συμμόρφωση των πελατών προς τα στάνταρ ISO πάντοτε μιλούσε για τελική διορία αλλά πολύ, ποτέ δεν μίλησε η υποχρέωση των πελατών να κάνουν κάτι οι ίδιοι. Υπάρχουν άλλες δυνατές λύσεις και κυρίως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές πληρωμών δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τους πελάτες να υποβάλουν τους φακέλους με βάση στάνταρ ISO και θα πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρξει νομική υποχρέωση για τους πελάτες και έχουμε ετοιμάσει σχετική διατύπωση. Για τις μελλοντικέ καινοτομίε, το παράρτημα που καλύπτει τις τεχνικές ε, προδιαγραφές θα πρέπει να συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται ενημέρωση κάθε ένα-δύο χρόνια, διότι οι αλλαγές στα συστήματα πληρωμών και οι βασικές τεχνικές αλλαγές χρειάζονται χρόνο και επίσης χρειάζεται μια βεβαιότητα για τους χρήστες στην αγορά να γνωρίζουν πώς ε, λειτουργεί κάτι στην πράξη. Αν δώσετε αυτή την εξουσία στην Κομισιόν και αποφασίσουν να αλλάξουν τα πράγματα κάθε χρόνο, θα δημιουργηθεί πρόβλημα θα δημιουργηθεί σύγχυση. Επίσης έχουμε κάνει και σε αυτό το σημείο σημαντική πρόοδο με την εισηγήτρια και θα επαναλάβω ότι ένα κοινό βήμα για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ας πούμε έτσι και τους χρήστες και τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς θα ήταν το Συμβούλιο ΣΕΠΑ για τη μεταβατική περίοδο. Είχε προτείνει δύο ε, προθεσμίες η Κομισιόν, μία για την μεταφορά πιστώσεων και την άλλη για την άμεση πίστοση. Νομίζουμε πως είναι σημαντικό να υπάρχουν δύο διαφορετικές τέτοιες ημερομηνίες, γι' αυτό προτείνουμε ε, μία ημερομηνία, μία προθεσμία αργότερα, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν τον αριθμό λογαριασμού και όλοι να έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν για το σημείο ε, ε, ε, συναλλαγής Νομίζω πως θα συζητηθεί περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Τραπεζών συμφωνεί με την θέση της Κεντρικής Τράπεζας και αναγνωρίζουν ότι το κόστος των ε, πολλαπλών συναλλαγών είναι μη ανταγωνιστικό σήμερα. Υπήρξε λοιπόν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αλλαγή του σχεδίου πρόταση με τρόπο που να οδηγήσει σε περισσότερη εναρμόνιση. Και εδώ το σημείο κλειδί είναι ότι η εναρμόνιση θα επιφέρει ανταγωνισμό. Αν παραμείνουμε στου εθνικού τρόπου ε, και επιμείνουμε πολύ, δεν θα έχουμε τον ανταγωνισμό που επιθυμούμε ανάμεσα στου προμηθευτέ και τα συστήματα. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Nous Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε αμέσως στην ε, κυρία για 7 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το χάρτη των μεταφραστών θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο αργά. Θα συντομεύσω λοιπόν την ε, παρουσίασή μου για να μείνω στα εντός του 7 λεπτού. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε που δίνετε την ευκαιρία στην ε, Όμιλο Κρεντή Αγκρικόλ να έρθει και να εκφράσει άποψη για ένα σχέδιο κανονισμού που μπορεί, αν ψηφιστεί ως έχει, να ανατρέψει εκβάθρων των ε, αγορά των πληρωμών στην Ευρώπη. Πριν να περάσουμε στην εξέταση των διατάξεων που μας ανησυχούν, θα ήθελα να θυμίσω κάποια αριθμούς κλειδιά της του μήλου μας. Είναι 54 εκατομμύρια ε, πελάτες στον κόσμο, πάνω από το μισό βρίσκονται στην Ευρώπη. Είναι ένας όμιλος ε, πολύ σταθερός, με ίδιους πόρους με, σε, της τάξης του 8,8%, αλλά είναι και μια, ένας συνεταιριστικός όμιλος με πάνω από 8 εκατομμύρια μετόχους, δηλαδή 8 εκατομμύρια πελάτες που είναι και μέτοχοί μας και που προσέχουν ιδιαίτερα τη διακυβέρνηση και την, ε, τις οικονομικές εξελίξεις. Έχουμε 7 δις ε, συναλλαγές ετησίως και ο όμιλός μας αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της αγοράς των πληρωμών στη Γαλλία και γύρω στο 5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το ε, σχέδιο κανονισμού, όπως ε, και οι συνάδελφοι συμφωνώ με αυτή την πρωτοβουλία γιατί θα επιτρέψει να πιστούν οι τελευταίοι διστακτικοί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να υιοθετήσουν ε, τις, τα εμβάσματα και την άμεση επίστοση ΣΕΠΑ που θυμίζω ετέθησαν στη διάθεση των πελατών τους πάνω από 5.000 τράπεζες στην Ευρώπη από το 2008 για τις, ε, τα εμβάσματα και από το 2009 για τις ε, αναλήψεις. Πρόκειται για καθολικές υπηρεσίες οι οποίες είναι διαλειτουργικές. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν θέλετε να μεταφέρετε, να εμβάσετε χρήματα προς έναν ε, ε, δικαιούχο το οποίο γνωρίζετε τις τραπεζικές, τα τραπεζικά στοιχεία δεν χρειάζεται καν να, ρωτηθεί, αναρωτηθείτε αν η τράπεζά σας θα μπορέσει να το κάνει. Είναι γενικώ παραδεκτό και εδώ ε, συμφωνώ με αυτά που είπε και η κυρία Βιλή ότι είναι δηλαδή βασικές υπηρεσίες και κανένας πελάτης μας δεν πρόκειται να ανησυχήσει να σκεφτεί αν αν θα πιστωθούν όντω τα χρήματα στο λογαριασμό του δικαιούχου και για έναν μεγάλο πιστωτή όταν αποφασίσει να, πάρει, να, να, σηκώσει αυτό που μπορεί από το λογαριασμό του δεν τον, δεν τον νοιάζει να ξέρει ακριβώς ποιος είναι, ποια είναι η τράπεζα που έχει το λογαριασμό του πελάτη του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ε, ε, στοιχεία για τη συνέχεια της συζήτησης. Και αυτό είναι δυνατόν διότι οι τράπεζες Ίσως να πω μια λέξη τώρα που δεν θα αρέσει πολύ στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, αλλά είναι γεγονός ότι οι τράπεζες συμφώνησαν να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες, να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και να χρησιμοποιήσουν τα ίδια στάνταρ, γιατί ανέπτυξαν συστήματα συναλλαγών και συντονισμού που επιτρέπουν να εκτελούν τις οδηγίες των πελατών τους με ένα επίπεδο ασφάλειας, επί του οποίου οι ποπτικές μας αρχές είναι εξαιρετικά ε, ε, ε, σε γρήγορση πάντα αυτό που μας ανησυχεί στο συγκεκριμένο κανονισμό είναι αυτή η ιδέα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληρωμών. Δεν θα έπρεπε για να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε στην, ε, στην ουσία ή να οθήσουμε για τη δημιουργία ε, ενό πανευρωπαϊκού συστήματος να υποχρεώσουμε ορισμένε τράπεζε, ορισμένε αγορέ να υλοποιήσουν επενδύσει που δεν αντιστοιχούν στι ανάγκε των πελατών του. Και θα σα δώσω το παράδειγμα τη ε, ανάληψη ενό σταθερού ποσού που δεν επιτρέπει στον πιστωτή να αρνηθεί ή να, ε, να αρνηθεί ή να ε, διαμαρτυρηθεί για μια τέτοια πίστοση. Η Τράπεζα της Γαλλίας πολύ επιφυλακτικά βλέπει αυτό το αυτή την πρόταση γιατί θεωρούμε πως δεν προχωρά προς το πνεύμα της οδηγίας αυτής αλλά ανοίγει ένα, ένα παράθυρο διαμαρτυρίας για τους ε, πιστωτές. Αυτό θα σήμαινε ότι όλες οι τράπεζες αυτού του είδους θα ήταν υποχρεωμένες να επενδύσουν για να μπορούν να λαμβάνουν αυτό, αυτές τις ε, πληρωμές, το reachability, του άρθρου 3.1, ενώ ο ίδιος τους ο πελάτης αρνείται αυτή την υπηρεσία. Και αν ε, ε, ε δεχόταν αυτή του είδους τη συναλλαγή θα ήταν υποχρεωμένη να την απορρίψει μαζικά. Πράγμα το οποίο θα καταστρέψει την εμπιστοσύνη που, πρέπει να, που οφείλουν να έχουν οι πελάτες μας σε ένα τραπεζικό σύστημα πληρωμών. Το... <coughs> Επίσης, άλλο πρόβλημα είναι αυτή η διάταξη για το οικονομικό πρότυπο και άρα η απαγόρευση προμηθειών ε, για τις συναλλαγές ε, και τις πληρωμές σε άμεση πίστοση. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν γιατί σε ορισμένες αγορές, ε, τις περίφημες έξι χώρες που αναφέρθηκαν, υπάρχει προμήθεια, ενώ σε άλλες όχι. Να σας πω ότι οι χώρες, οι έξι, όπου υπάρχει προμήθεια για την άμεση πίστοση, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60%, 70% των ε, αναλήψεων που γίνονται στην Ευρώπη. Και στις άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει αυτή η προμήθεια, μετά από την εφαρμογή της άμεσης πίστοσης, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2009, ε, δεν έχει διαπιστωθεί κίνηση, μαζική κίνηση μεταφο... μετάβαση σε αυτό το σύστημα, ούτε και σε αυτές τις αγορές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να πούμε ότι το σύστημα βασίζεται ε, μάλλον οικοδομείται με τον καιρό, είναι πολύ ευαίσθητο το να αλλάξει ξαφνικά το οικονομικό πρότυπο γιατί μπορεί αυτό να αποσταθεροποιήσει την αγορά. Και γι' αυτό και πιστεύω πως σήμερα η πρώτη πρόταση της, της εισηγήτριας της κυρίας είναι πολύ ενθαρρυντική και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το διάλογο ακριβώς έτσι ώστε να εξελιχθεί το κείμενο, να, υπάρξει, να είναι πιο αποτελεσματικό για όλους. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, είστε καταπληκτικοί. Επτά λεπτά και τρία δεύτερα. Euh, ο κύριος Έπινγκ, ο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Φέρμπερ μετά. Ο κύριος Σέπινγκ, ευχαριστώ. Στα αγγλικά ο κύριος Σέπινγκ. Έχω μερικές ερωτήσεις για αυτά τα θέματα. Μετά ε, από τις ομιλίες που ενέκυψαν διάφορα προβλήματα και το ένα είναι το IMF, ε, η πολυμερή τέλη συναλλαγών. Και είναι ένα θέμα αναλογικότητας. Γιατί ένα έμβασμα κοστίζει λεφτά και γι' αυτό υπάρχει και τέλος. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν, ε, ούτε δωρεάν γεύματα για μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια προσέγγιση, ε, Dot Frank στις Ηνωμένε Πολιτείε, είναι μια νομοθεσία του πρώην γερουσιαστή Κρίς Dot και του βουλευτή ε, στη Βουλή των Αντιπροσώπων του κυρίου Φρανκ. Ε, και θα πρέπει να μας εμπνεύσει. Βασίζεται σε ένα χαμηλό τέλος και αν υπάρχουν υψηλότερα έξοδα να αποδεικνύεται αυτό. Εγώ δεν αποκλείω αυτό λοιπόν να μην υπάρχει κανένα τέλος γιατί θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιο κόστος. Και το δεύτερο είναι η τελική ημερομηνία. Και έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Χάστινγκ. Βεβαίω, η καταληκτική ημερομηνία είναι κάτι σημαντικό γιατί βοηθάει να προχωρούν τα πράγματα και περιμένει και αγορά, ξέρει μάλλον τι την περιμένει, συγγνώμη, και κανονίζει την πορεία τη. Και είναι και πιο αποτελεσματική. Ε, με μια συντονισμένη μετάβαση ε, στο σύστημα από αυτό που ισχύει σήμερα των ε, κρατικών ε, εθνικών εμβασμάτων στα άλλα ευρωπαϊκά. Λέει η κυρία Βίγκε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε άλλες χώρες και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χάστινγκ ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχετε στο μυαλό σας. Προθεσμία, ημερομηνία και έτος. Και έχω και μια ερώτηση για τις εξαιρέσεις προς την κυρία Βαντχιόβερ. Ξέρουμε ότι στη Γερμανία υπάρχει η ε, ηλεκτρονική διαδικασία εμβασμάτων διαφορετική από τη διαδικασία IBAN. Και τι θα γίνει τώρα. Θα Πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα περιορισμοί, γιατί η Γερμανία είναι μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς και να έχουν ήδη τόσες μεγάλες εξαιρέσεις ε, είναι αντίθετο προς την ιδέα ε, μιας πανευρωπαϊκής ε, ζώνης ή χώρου πληρωμών. Αυτά είχα να ρωτήσω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μα μπορώ που τα ξέρει τόσο καλά τα γερμανικά προβλήματα ο κύριος Σέπινγκ, μου πήρε την ερώτηση από το στόμα. Ήτανε, ήτανε και στο γραφείο του Επιτρόπου Μπόλκενστάιν και τα ξέρει ε, αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τα βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα το έμβασμα. Ξέρετε πως ε, πρέπει να λυθεί το ζήτημα των ε, εξουσιοδοτήσεων για την ανάληψη από το λογαριασμό και βέβαια και το ζήτημα το οποίο ανέφερε ο κύριο Σέπινγκ για το σύστημα που έχουμε στη Γερμανία το οποίο βεβαίως ε, θα αντικατασταθεί αν τεθεί το ΣΕΠΑ και θα πρέπει να αλλάξει τελείως το σύστημα και βεβαίως ε, θα ακολουθούν θα καταργηθούν άλλα συστήματα που υπάρχουν ήδη. Αντιλαμβάνομαι τις τράπεζες που θέλουν μόνο ένα σύστημα, να έχουν δηλαδή παντού το ΣΕΠΑ. Το καταλαβαίνω λίγο, αλλά ε, δεν μπορεί αυτό να κανονίζει το πώς θα είναι τα, τα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει το ΣΕΠΑ ως ένα μίνιμουμ και επιπλέον να συνεχίσουν να υπάρχουν ε, οι... τα υπόλοιπα συστήματα. Επίσης θα μιλάμε για αυτό το βιβλίο των κανόνων σε αντίθεση με μια οριστική ημερομηνία ε, φαίνεται πως ε, σε εκείνη την ημερομηνία θα, θα εξαφανιστούν πάρα πολλές ε, υπηρεσίες γιατί δεν προβλέπονται στο ΣΕΠΑ. Θα μπορούσε λοιπόν να διασφαλιστεί μια παράλληλη ύπαρξη αυτών των συστημάτων και μετά από αυτή την τελική ημερομηνία. Η συγκήτρια θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Φίλη που εκπροσωπεί τους καταναλωτές. Πώς βλέπετε το ρόλο του Συμβουλίου της ΣΕΠΑ. Είπατε κάτι γι' αυτό, αλλά ε, πώς ε, προτείνετε να βελτιωθεί αυτό. Δεν είναι ικανοποιητικό, λέτε αυτή τη στιγμή. Πώς βελτιώνετε, τι προτείνετε εσείς για να είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές και να ακούγεται τη φωνή τους καλύτερα. Επίσης υπάρχουν πολλές ρήτρε για την προστασία των καταναλωτών στο κείμενο αυτό του κανονισμού. Σας ικανοποιούν. Εκεί βλέπετε κανένα περιθώριο βελτίωσης. Ιδιαίτερα ε, όταν πρόκειται για την ασφάλεια των συναλλαγών. Και μια τρίτη ερώτηση. Τι είδους ενημερωτικές εκστρατείες και βοήθεια περιμένετε από τις τράπεζες για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές. Πώς θα πρέπει ή πώς μπορεί να βοηθήσει πάση περιπτώσει ο τραπεζικός τομέας για να φτάσει η πληροφόρηση ε, στους καταναλωτές για τις αλλαγές που χρειάζονται για τις πληρωμές στο χώρο ΣΕΠΑ. Και κύριε Χάρτσινγκ, παρακαλούσα, θέλετε να απαντήσετε κι εσείς σε αυτό το τελευταίο ερώτημα. Είναι έτοιμος ο τραπεζικός τομέας να υποστηρίξει κάπως. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, για όλους μας ο τραπεζικός μας λογαριασμός είναι πολύ ευαίσθητη υπόθεση και θέλουμε να ξέρουμε τι αλλαγές υπάρχουν, αλλαγές στις πληρωμές, πώς θα ενημερωθούμε για αυτές και πώς θα ενημερώσουμε τους καταναλωτές μας. Επίσης θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χάρτσινγκ. Εγώ άκουγα τη μητρική μου γλώσσα τη μετάφραση στα φιλανδικά. Δεν ξέρω αν είπατε. Θέλετε να α, ε, απαλληφθεί τελείως το άρθρο 6 ή ήταν καμία παρεξήγηση. Ε, που θέλετε να το αναθεωρήσετε, ε, να το τροποποιήσετε ή τι θέλετε να το καταργήσετε τελείως. Και πώς θα υπάρχουν οι κανόνες παιχνιδιού διαφορετικά για όλες τις τράπεζες σε διάφορα κράτη-μέλη και τις συναλλαγές και τα τέλη της προμήθειας συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, τα διατραπεζικά αν τελείως καταργηθεί. Ε, merci Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής μας. Αν όχι, θα δώσω τότε το λόγο πρώτα στον κύριο Χάρτσεν για να απαντήσει, γιατί σας έκανα πολλές ερωτήσεις και άμεσες και μετά στους υπολείπους. Και επίσης, επισημάνω ότι παρευρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσουμε και σε εκείνους το λόγο, αν το επιθυμούν, ή πριν απαντήσουν. Αν θέλετε να μιλήσετε τώρα, να το πείτε. Ο κύριος Χάρτσεν όμως πρώτος. Νομίζω πως ήταν ε, και μια ερώτηση για την ε, κυρία Φιλή. Για την ε, τελική ημερομηνία η θέση της EPC ήταν σαφής. Πάντα λέγαμε πως ναι πρέπει να υπάρχει μια τελική ημερομηνία. Γι' αυτό το λόγο καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του ΕΚΟΦΗΝ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δίνουν εντολή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει μια πρόταση για μια τελική ημερομηνία. Το θέμα και το ερώτημα ήταν ποια είναι αυτή η τελεία ημερομηνία. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών είπαμε πω θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ημερομηνία οριστική για όλη την Ευρωζώνη και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τι χώρε εκτό Ευρωζώνη το τι θα κάνουμε, ειδικά με αυτές οι οποίες ε, ίσως σε γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Οπότε κάνουμε μια διάκριση μεταξύ Ευρωζώνης και λοιπόν ε, αγορών στα κράτη-μέλη. Δεν τοποθετηθήκαμε για την ε, τελική αυτή ημερομηνία, αλλά ίσως θα έπρεπε να υπενθυμίσω σε όσους παρακολουθούν το τι κάνουμε. Ιστορικά λέμε Πώς? Εργαζόμαστε πάνω σε ένα μοντέλο για να είμαστε έτοιμοι να το υιοθετήσουμε και ξέρετε πως τελικά η οδηγία πληρωμών καθυστέρησε τουλάχιστον δύο χρόνια και άρα στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπανε το Μάρτιο του 2009 και 2010 πως θα πρέπει η τελική ημερομηνία να είναι το Μάρτιο 2012. Είμαστε τώρα στο 2011 και ακόμα δεν έχουμε τελική θέση για το ποια θα πρέπει να είναι η τελική ημερομηνία αλλά παρατηρούμε πως υπάρχουν δύο τελικές ημερομηνίες που αναφέρονται. Δεν μας αρέσει αυτό. Εμείς προτιμάμε όπως είπα μία. Οπότε, αν ε, το Κοινοβούλιο έχει μια συγκεκριμένη ε, πρόταση, θα επανέλθουμε κι εμείς ε, στην συνέλευση των μελών μας. Υπήρξε επίσης ένα ερώτημα του εισηγητή για το πώς θα διαχειριστούμε τις άλλαγες και το θέμα του Συμβουλίου της ΣΕΠΑ. εξ ονόματος νομίζω των συναδέλφων μου, ξεκαθάρισα πως εάν δοθεί εξουσία μόνο μερός στην Κομισιόν, ε, δεν είναι σωστό ε, μοντέλο αυτό και άκουσα προσεκτικά ε, κυρία η οποία μίλησε πριν από λίγο και Βεβαίω ε, την κυρία Τούμπελ Κουκερέλ και αν χρειαστούν πάρα πολλέ αλλαγές και αλλάξουν οι ε, αγώνες, οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν μόνο για τους συμμετέχοντες στο σύστημα και όχι για τους πελάτες. Τεχνικές προδιαγραφές επίσης ισχύουν ε, και για τους πελάτες. Αλλά έχει κάποιο νόημα νομίζω να ζητήσουμε στο τέλος συμβουλές και από την Κεντρική Τράπεζα και το είπα πως το άρθρο 22 του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δίνει στην στο σύστημα, το ευρωσύστημα την δυνατότητα να ορίσει προδιαγραφές. Αλλά αυτό είναι μόνο για τις συναλλαγές ε, μεταξύ τραπεζών. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να ζητήσουμε μια σύσταση στο Συμβούλιο ε, ΣΕΠΑ όπου βεβαίως ε, συμμετέχουν και οι πρόεδροι του EPC και των πελατών και της δημόσιας διοίκησης. Οπότε αυτοί λένε το εάν θα πρέπει να εφαρμοστεί μια τεχνική προδιαγραφή. Αυτό το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως οι τεχνικές προδιαγραφές, εάν αλλάξουν δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις τράπεζες, όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι δημόσιες διοικήσεις και τεχνική, υπάρχει τεχνικών λύσεων ε, πρέπει να αλλάξουν. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης για τα χαρακτηριστικά αυτά τα προαιρετικά για τις, ε, άμεσ, για τις ε, άμεσες εντολές ε, πληρωμής 8 εβδομάδων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε περισσότερα από αυτά τα οποία ορίζει η οδηγία. Έχουμε μια περίοδο 8 εβδομάδων εντός των οποίων θα λάβουν πίσω τα λεφτά οι πελάτες χωρίς πολλά πολλά. Και αν μια δημόσια διοίκηση ή κάποια επιχείρηση κάνει κατάχρηση αυτής της εντολής με το να ξεκινήσει μια τέτοια χρέωση και ε, αυτό δεν είναι σωστό, έχει τουλάχιστον ένα έτος για να λάβει τα λεφτά του πίσω ο καταναλωτής. Οπότε ακόμα και αν δεν γίνει εντός της ε, περίοδου αυτής. Εάν λοιπόν ταυτόχρονα γίνει υποχρεωτικό από πλευράς νομοθεσίας πως ε, για κάθε πληρωμή πρέπει να γίνει έλεγχος, τότε θα δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ακριβό σύστημα πληρωμών στην Ευρώπη που δεν χρειάζεται. Γιατί ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα ούτως ή άλλως να πάρει τα λεφτά του πίσω. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φιλή. Θέλετε να απαντήσετε πριν... Oui, c'est bon. <laughs> Merci, madame. Alors, en ce qui concerne la première... Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση για τα τέλη και ότι τίποτα δεν είναι στη ζωή δωρεάν και πρέπει να την υπόψη το κόστος. Εντάξει, το ξέρω αυτό, αλλά δεν νομίζω να είπα εγώ να είναι τελείως δωρεάν ε, ε, η ε, πράξη αυτή, η συναλλαγή. Επανειλημμένα ακούσαμε ότι σε έξι χώρες υπάρχει αυτό το σύστημα IMF των πολυμερών τελών. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι το πληρώνουν ε, οι ε, καταναλωτές. Εγώ πληρώνω κάθε χρόνο στην τράπεζά μου προμήθειες και μπορούν να ζητήσουν για κάθε νέα ε, πάγια εντολή που δίδεται να πληρώνει κάποιο ποσό σύμφωνα με την πράξη και τη συναλλαγή κάθε φορά. Θα μπορούσε να ασχοληθεί κανείς ε, σοβαρά με αυτό το θέμα της χρέωσης ανασυναλλαγή με βάση του πραγματικού κόστους έτσι και όχι πολύ υψηλά ε, τέλη με τον όρο και την προϋπόθεση μόνο να γίνονται έλεγχοι, επαληθεύσεις ε, και από το κράτος και μάλιστα τακτικά ως προς το ύψος των τελών που ε, χρεώνουν οι τράπεζες και από εκεί και πέρα να μην πληρώνουν επιπλέον οι καταναλωτές. Δεν μπορούν να έχουν αυτά τα τέλη και άλλες προμήθειες. Ε, όπως λέμε σε μια παροιμία, ας πούμε, λέει ότι δεν μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Επίσης, οι καταναλωτές δεν είναι οι πρώτοι ε, εποφελούμενοι ε, αυτής της ε, υπηρεσίας. Οι δικαιούχοι είναι εκείνοι που παίρνουν τα χρήματα, όχι αυτός που στέλνει το έμβασμα. Και όταν γίνεται αυτόματη πληρωμή από ένα λογαριασμό σε άλλο, να υπάρχει κάποιο λογικό τέλος, αλλά όχι υπερβολικό. Τώρα για το Συμβούλιο ΣΕΠΑ. Ως καταναλωτές συζητήσαμε και ζητήσαμε και με άλλους ε, ενδιαφερόμενους και χρήστες να δημιουργηθεί αυτό το Συμβούλιο ΣΕΠΑ για να υπάρχει ε, ένα ουδέτερο όργανο όπου θα συνεδριάζουν όλα τα ενεχόμενα μέρη. Θελήσαμε αυτό το Συμβούλιο να έχει ένα ρόλο διαιτητικό. Αυτό μας το αρνήθηκε το ίδιο το Συμβούλιο. Ε, εκτός αυτού, όπως είπα και στην αρχή, είναι σημαντικό για μας επίσης να σκεφτούμε έναν άλλον οργανισμό που να αποφασίζει για τους τεχνικούς κανόνες. Δεν μπορεί να είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών που θα ορίζει τους κανόνες, γιατί είναι μόνο ένα τμήμα της αγοράς αυτό. Δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χρηστών, τα οποία μετράνε πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τη ρήτρα προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο κανονισμού χωράνε και οι βελτιώσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί οι κανόνες που σήμερα περιλαμβάνονται στο κείμενο, ε, όλους αυτούς είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν και δεν εισακούστηκαν τότε τα αιτήματά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επανέρχεται στη βαρούσα πρόταση κανονισμού. Και βέβαια υπάρχουν σημεία που θέλουμε να βελτιώσουμε η προμήθεια που θα πληρώνει ο καταναλωτής ας πούμε σε περίπτωση απόρριψης μιας πληρωμής να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει μόνο σε περίπτωση που δεν έχει αρκετά χρήματα στο λογαριασμό του τη στιγμή που πρέπει να καταβληθεί αυτή η πληρωμή λόγω της πάγιας εντολής. Δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο σε περίπτωση απόρριψης να πληρώνει και ο καταναλωτής. Και σε ό,τι αφορά ένα ποσό συγκεκριμένο κάθε φορά, και εδώ χρειάζεται βελτίωση χωρίς να το ζητούμε εμείς βέβαια να υπάρχουν κανόνες ειδικοί, αλλά σε περίπτωση που μπει κάτι στη ε, οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών θα πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα οι καταναλωτές όταν έχουμε πάγιες εντολές με σταθερά ποσά κάθε φορά. Ε, το άλλο θέμα, οι ενημερωτικές εκστρατείες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε ε, σε ένα συμβούλιο, σε μια συνεδρία του Συμβουλίου της ΕΠΑ και εμείς ως εκπρόσωποι των καταναλωτών τοποθετηθήκαμε όπως και άλλοι και είμαστε υπέρ και παραμένουμε μια ε, ε, μιας ενημερωτικής τύπου σαν αυτή που χρησιμοποίησαμε δηλαδή για το ευρώ. Το ξέρετε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί καταναλωτές που δεν έχουν ακούσει τη ζωή τους στην ΣΕΠΑ και έχει ρόλο εδώ να διαδραματίσει και το δημόσιο. Βεβαίως και εκείνοι που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα ε, ενημερωτικά, αλλά και ως μέσον ότι κοιτάξτε υπάρχει αυτό το εργαλείο. Το Άιμπαν στη Γερμανία το λένε τώρα Ιβάνο Τρομερός το έχουν βαφτίσει. Ε, και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα μετατροπής των εθνικών συστημάτων, σε ένα, στο σύστημα IBAN, τα ξέρετε αυτά, σε διάφορες χώρες που διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών. Και ένα τελευταίο, μεταβατικές περίοδοι για κάποια ειδικά προϊόντα. Εδώ γίνεται λόγος για κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολύ τους Γερμανούς. Από μια χρεωστική κάρτα να, γίνονται, να δίνονται εντολές τέτοιες, αυτό ικανοποιεί πάρα πολύ τους Γερμανούς καταναλωτές και δεν θα πρέπει να καταργηθεί. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο χώρος ΕΠΑ να είναι η ευκαιρία να προβληθεί αυτό και αλλού στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίγκε έχει το λόγο. Άμα επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση των ε, διατραπεζικών συναλλαγών. Πάντα αυτό ταυτίζεται με ένα τέλος που επιβαρύνει άμεσα τον καταναλωτή, γιατί όλοι εκινούν από την αρχή ότι ο έμπορος ας πούμε ή ο πιστωτής ε, μετακυλεί το κόστος στον καταναλωτή. Επίσης κατηγορείται το σύστημα αυτό για διαφάνεια. Θα ήθελα να θυμίσω το ποσό που διακινείται με αυτόν τον τρόπο. Είναι ε, δημοσίως γνωστό. Επίσης, ε, στο κόστος που συναπαρτίζει την τιμή των εμπόρων και των πιστωτών λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα πληρωμών. Εμείς ας πούμε δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει ε, όταν πληρώνεται σε μετρητά ο, ο έμπορος, ούτε πώς κοστολογεί ε, το τελικό του προϊόν ο έμπορος με βάση τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώσω. Όταν μπαίνω σε ένα μαγαζί ε, δεν ξέρει αν θα τον πληρώσω με επιταγή, ε, με κάρτα ή με μετρητά. Τα IMF αυτά τα τέλη δεν είναι άμεση επιβάρυνση της τιμής του τελικού καταναλωτή. Συνυπολογίζεται βεβαίως ένα μείγμα σε ένα κόστος και σε έναν υπολογισμό που ακολουθεί ο έμπορος για να καθορίσει την τελική τιμή του προϊόντος. Όταν μας λέτε ότι τα τέλεια είναι πολύ ακριβά, αυτό πώς ορίζεται, ωραία, και πώς υπολογίζεται τι κοστίζει ε, η ίσπραξη μιας επιταγής ή με κάρτα ή με μετρητά. Ε, δεν είναι ακριβώς ταυτόσημα όλα αυτά τα μεγέθη. Και επίσης αν διατηρηθεί αυτό το σύστημα διασυναλλαγών, ε, κάποιοι λέγουν ότι αυτό σημαίνει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το αντίθετο, αν καταργηθούν θα είναι τεράστια η στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ε, τραπεζών των ε, πιστωτών που είναι λίγες, ενώ είναι πάρα πολλές οι τράπεζες εκείνων που πληρώνουν που πρέπει να κάνουν τις επενδύσεις για να μπορούν να δέχονται αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή, σε ένα σύστημα πάγιας εντολής πληρωμής θα πρέπει να στηθεί αυτό το σύστημα ε, για να ε, μπορεί η τράπεζα να τα αποκρίνεται. Ενώ εκείνοι που πληρώνουν, οι μεγάλες εταιρείες ε, είναι πελάτες κάποιων τραπεζών και μόνο. η City Group, ο Όμιλος, ας πούμε, είναι μια μεγάλη τράπεζα που εργάζεται η παρακαθήμενη. Ε, για μένα το να απαγορευτεί αυτές, αυτή η μορφή της είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ακριβώς τρέβλωση του ανταγωνισμού. Γιατί επιβαρύνονται οι τράπεζες οι οποίες θα πρέπει να στήσουν αυτό το σύστημα. Αν αρχίσουμε, κινήσουμε από την αρχή που λέγει ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν να πληρώνουν περισσότερο και θα πρέπει περισσότερο οι τράπεζες τους να επενδύουν και αν καταργηθεί και αυτό το σύστημα αποζημίωσης δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα συνολικά και πώς θα χρηματοδοτείται ή οι τράπεζες των ΜΕ θα χρηματοδοτούν τις τράπεζες των ΔΕ. Ευχαριστώ. Έχουμε πρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που μπορεί να σας απαντήσει. Θα δώσω όμως το λόγο στην κυρία Βαντφέφερ πρώτα για να απαντήσει σε ερώτηση που έγινε. Okay, um, I would like to just make two points. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο αφορά ένα ερώτημα του κυρίου Έπινγκ και το ανέφερε και ο κύριος Φέρμπερ. Νομίζω πως η ΣΕΠΑ είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και στόχο έχει να φέρει ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι εθνικά συστήματα, κανόνες. Έχουμε σε κάποιες χώρες διάφορα, <coughs> διάφορα συστήματα, αναφέρθηκε το γερμανικό σύστημα που διαφέρει από τη χρέωση της ε, ΣΕΠΑ και σε άλλες χώρες και έχουμε και την κανονική χρέωση συν ε, το έμβασμα στην Γερμανία. Οπότε πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τι υπάρχει σε κάθε χώρα. Ήδη δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς αυτό, αλλά ξέρουμε πως υπάρχουν κάποια μεγάλα συστήματα, όπως το γερμανικό ή το ρίμπα της Ιταλίας, που ε, λειτουργούν κάπως διαφορετικά, όσον αφορά δηλαδή την εμπειρία του πελάτη. Μετά το δεύτερο ερώτημα είναι πως θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτά τα συστήματα ενώ περνάμε σε ένα ενιαίο πρότυπο για την επεξεργασία γιατί βεβαίως το ΣΕΠΑ είναι πρότυπο οπότε αυτό δεν σημαίνει πως ο πελάτης ε, θα έχει το ίδιο προϊόν σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ευρώπη, θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικά επίπεδα, διαφορετική τιμή ανάλογα του εάν προσφέρεται μέσω κινητού τηλεφώνου, χαρτιού ή μέσω διαδικτύου, γιατί όλα αυτά βεβαίως είναι και θέματα ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. Οπότε, Μπορεί κάποια συστήματα να φύγουν τελείω από την αγορά, αλλά κάποια μεγάλα αλλά θα πρέπει να τα εξετάσουμε να δούμε πώς θα αλλάξουν. Στις συναλλαγέ ε, του γερμανικού συστήματος υπάρχει ένα συνδυασμό ε, χρέωσης ε, που λαμβάνει χώρα μεταξύ των τραπεζών και ο έμπορος διαβάζει την κάρτα του πελάτη και υπογράφει ο πελάτης ένα χαρτί για να ξεκινήσει κατ' ουσίαν ένα σύστημα χρέωσης. Ένα ευρετικό δηλαδή σύστημα λειτουργεί στη Γερμανία γιατί στη Γερμανία ο κόσμος πληρώνει αυτό το οποίο θέλει να αγοράσει και άρα δεν χρειάζονται μια συναλλαγή με εγγύηση της τράπεζας. Δεν βασίζεται λοιπόν σε κάποια κάρτα, κάποια Visa, Mastercard ή κάποια άλλη. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησαν οι έμποροι και οι έμποροι μετά αναλαμβάνουν τον κίνδυνο του εάν θα πληρώσει ο πελάτης ή όχι. Έχουμε και άλλα συστήματα σε άλλες χώρες που λειτουργούν κάπως διαφορετικά και αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο είναι να δούμε ποια από αυτά τα συστήματα υπάρχουν, ποια είναι μεγάλα και να δώσουμε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Ξέρω πως το Κοινοβούλιο πρότεινε το 2015 για τα μεγαλύτερα αυτά συστήματα που συνεπάρχουν μαζί με το ΣΕΠΑ. Το Συμβούλιο μπορεί να δώσει και άλλο ένα έτος, οπότε θα έχουμε μία περίοδο προσαρμογής ή κατάργησης του συστήματος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι πελάτες αμέσως θα δουν επιδείνωση των υπηρεσιών τους. Μετά, κατόπιν, ε, αυτό το οποίο είναι πρόκληση για τον ε, κλάδο είναι το πώς θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός μεταξύ των ε, τραπεζών γιατί σήμερα κρύβονται πίσω από εθνικές προδιαγραφές και συστήματα οπότε υπήρξε κάποια εναρμόνιση αλλά τώρα πλέπει βεβαίως ε, και το κοινό να το αγκαλιάσει και οι ιδιώτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν σαν ομοσπονδιακή κυβέρνηση να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες του κλάδου γιατί βεβαίως αυτά γίνονται για τον ανταγωνισμό, δεν ε, θα μειωθεί ο ανταγωνισμός έτσι των τραπεζών και, να, και θα εκμεταλλευτούν τους, τους χρήστες, θα ανοίξουν την αγορά και θα έχει την επιλογή ε, ο πελάτης μεταξύ μιας γαλλικής τράπεζας, μιας φιλανδικής τράπεζας ή ενός άλλου ιδρύματος που δεν θα είναι τράπεζα. Οπότε θα πρέπει να το δούμε ως, από την πλευρά του κλάδου, του χρήστη και της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Έγινε πολλής λόγος για ανταγωνισμό. Και από πλευρά τη κυρία Βιγκέ που δεν θέλει στρέβλωση και αφού έχουμε τη χαρά να έχουμε μεταξύ μας την κυρία Ρίτα Βέζεμπεκ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ανταγωνισμού, της δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε και αν αυτή ήταν η ερώτησή σας, θα ήθελα να αναφέρω διάφορα πατρίσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό που έγιναν. Καταρχήν όσον αφορά την αναλογικότητα του κανονισμού. Νομίζω η Κομισιόν πιστεύει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και ότι η ρύθμιση των ε, προμηθειών είναι απαραίτητη και αναλογική. Ούτε η νομική υπηρεσία της Επικομισιόν, ούτε η οικονομική υπηρεσία του Συμβουλίου διαπίστωσε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, ο λόγος για τη ρύθμιση ε, των IMF σε αυτό το κανονισμό είναι ότι η ιστορία, της ε, το ιστορικό μάλλον της συζήτηση είναι ότι οι αντιρρήσεις της αλλαγής των τελών αυτών από την άποψη της, του ανταγωνισμού αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για τις, την μετάβαση των τραπεζών οι Τράπεζε διαμαρτύρονται ότι δημιουργείται έλλειψη σαφήνεια και κατά την άποψή του δημιουργείται και έλλειψη ισότιμου πεδίου ε, και καθιστά δύσκολη την κίνηση των τραπεζών. Εμείς από την άποψη της ΓΔ Ταγωνισμού θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων ε, μεμονωμένα και η αναπερίπτωση αξιολόγηση είναι ο κανόνας. Όμως, εφόσον εδώ πρόκειται για ένα δίκτυο, μια αγορά με δίκτυο, θα πρέπει να έχουμε ένα επαρκή αριθμό τραπεζών που θα κινηθούν στο σύστημα αυτό. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, θεωρούμε πως είναι καλύτερο σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση να ρυθμίσουμε αυτό που θα πρέπει να ισχύει σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού. Η λύση που επιλέξαμε είναι να περιγράψουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θα προκύψει από μια αξιολόγηση από τον ανταγωνισμού. Ε, το δεύτερο ζήτημα που επίσης ανέφερε η ΠΣ είναι γιατί αυτός ο κανονισμός να επεκτείνεται σε διμερείς και μονομερείς συμφωνίες. Διότι σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού η εκτίμηση των μονομερών και διμερών συμφωνιών είναι διαφορετική. Το άρθρο 6 όμως ε, έχει μπει εδώ ακριβώς ε, από, μέσα σε μια νομοθετική προσέγγιση και με την βούληση να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πεδίο για όλους. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό έχει νόημα να ασχοληθούμε και με τα άλλα είδη προμηθειών και να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει μια μειόμορφη ρύθμιση. Τώρα, πέρα από το να υπάρχει μία προμήθεια ή ε, διάφορες προμήθειες έχουν υποθεί πολλά. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει διαφορά σε μια αξιολόγηση ανταγωνισμού ανάμεσα στις προμήθειες που είναι κρυφ και που σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν το σύνολο του συστήματος και επιβάλλονται ε, επί τη βάση κάθε συναλλαγής ή της ε, προμήθειας που επιβάλλουμε εμείς ανά συναλλαγή, πιστεύουμε ότι για τις κρυφές προμήθειες που επιβάλλονται ένα συναλλαγή δεν βλέπουμε λόγο ύπαρξης. Η δικαιολόγηση τέτοιων προμηθειών εν γέννη είναι ότι οι κοινοφελείς υπηρεσίες έχουν συμφέρον να βάλουν τους καταναλωτές να πληρώσουν αυτό το πολύ ε, αποτελεσματικό τρόπο και θέλουν να επιδοτήσουν κατά κάποιο τρόπο το καταναλωτό. Καταναλωτή. Βέβαια, αυτές οι εταιρείε μπορούν να το κάνουν μόνος, μπορούν να κάνουν κάποια έκπτωση για να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής αυτήν αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο πληρωμής και δεν χρειάζεται οι τράπεζες να έχουν δικό τους μηχανισμό ε, επιδότησης. Αυτό είναι για τις προμήθειες ανά συναλλαγή. Τώρα, για τη δική μας, για τη δική μας πρόταση είναι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με κοινή συμφωνία θέλουν να επιβαρύνουν το, με το κόστος που προκαλείται από τα σφάλματα να επιβαρύνει το μέρος που έχει διαπράξει το σφάλμα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πείσεις κάποιον να πληρώσει επειδή κάποιος άλλος έκανε λάθος. Έχει νόημα λοιπόν να υπάρχει μια συλλογική ρύθμιση γι' αυτά. Ε, τώρα, για τις γαλλικές τράπεζες που λένε ότι τα, οι προμήθειες είναι δημοσιευμένες και ότι είναι γνωστές σε όλους, ε, από την εμπειρία μας να σας πω ότι δεν τα βρίσκουμε στα site των τραπεζών, δεν τις έχουμε λέξει βέβαια και όλες, αλλά εν γέννη δεν κυκλοφορούν και σίγουρα δεν ισχύει ότι αν εγώ ως καταναλωτής μπω σε μια ρύθμιση άμεσης επίστοσης, ότι ενημερώνομαι εκ των προτέρων ε, ότι θα γνωρίζω ότι κάθε φορά που κάνω μια πληρωμή το, το αντίθετο μέρος, ε, συνήθως δηλαδή η εταιρεία ηλεκτρισμού ή νερού κτλ. δεν το ξέρει ότι εγώ υποχρεώμαι να καταβάλω ένα τέλος, μια προμήθεια. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένε τράπεζες που, που, εξαρτώνται πολύ στο επιχειρηματικό του μοντέλο από τι προμήθειε και είναι οι τράπεζε καταναλωτικέ αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι είναι μια εξαιρετική κατάσταση όπου οι τράπεζες μόνο βοηθούν τους καταναλωτές. Ο κανονική κατάσταση είναι να υπάρχουν καταναλωτικές τράπεζες που, αλλά που συνήθως βοηθούν και τους καταναλωτές και ε, εξυπηρετούν μάλλον και καταναλωτές και επιχειρήσει. Υπάρχουν λίγες ε, περιπτώσεις ε, τραπεζών που βασίζονται στα έσοδα λόγω αυτών των κρυφών ε, τελών που επιβάλλουν κάθε φορά που ένας καταναλωτής κάνει μια πληρωμή. Είναι πολύ εύκολη η ροή εσόδων αυτή και οι τράπεζες φυσικά και θέλουν να τα τηρήσουν. Αλλά είναι μια πολύ μειοψηφία τραπεζών σε λίγα κατημέλια και δεν πιστεύουμε πως το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές θα πρέπει να καθοριστεί από αυτή τη μικρή μειονότητα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Απτά. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι η κυρία Βεγγέ δεν συμφωνεί καθόλου με αυτά που λέτε. Η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, έχετε και εσείς το δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας μετά από τη σφόδρη κριτική. Αν μου επιτρέψετε όμως να δώσω το λόγο σύντομα στην κυρία Βεγγέ και στον κύριο Χάρτσινγκ για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ε, κύριε Βιγκέ, εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά να πω το εξή. Να σας εκθέσω ποια είναι η πραγματικότητα. Αν θεωρήσουμε τη γαλλική αγορά, την οποία γνωρίζω καλύτερα βεβαίως από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, 20 μεγαλύτεροι ε, πιστωτές ε, εκπροσωπούν 80% ε, των εμβασμάτων που γίνονται από λογαριασμούς των πελατών. Αν δείτε, στις μεγάλες τράπεζες αυτό μοιράζεται ε, βέβαια, ε, αλλά αν το επιμερίσετε σε λεπτομέρειες, στην Credit Agricole έχουμε 39 περιφερειακά ταμιευτήρια που είναι αυτόνομες τράπεζες και είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από τράπεζα σε τράπεζα. Δηλαδή, όλες αυτές οι τράπεζες έχουν το ίδιο επίπεδο επενδύσεων να κάνουν και όταν δεν έχουν την τύχη να έχουν πελάτες αρκετούς ε, από ε, πιστωτές ε, για να εξισορροπήσουν την κατάσταση βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση σε περίπτωση που καταργηθούν τα τέλη γιατί χρειάστηκε να κάνουν την ίδια επένδυση με τους υπολείπους. Έτσι. Euh, Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και όπως συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκεί δηλαδή οι πιστωτές να προτείνουν στους πελάτες τους εκτόσεις, rebate, για την άμεση χρέωση, αν αυτό θέλουν να πληρώσουν με άμεση χρεωστική κάρτα. Ορισμένοι από αυτούς λοιπόν, αντί να προτείνουν ε, στους πελάτες πλεονεκτήματα, επιβαρύνουν ε, άλλο τρόπο πληρωμής, ενώ αυτό υποτίθεται ότι απαγορεύεται στη Γαλλία μετά τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ελέγξεις τον πιστωτή. Τι θα προτείνει στον πελάτη. Αν θα του προτείνει πλέον εκτήματα ή αν θα τον επιβαρύνει και με ένα χαράτσι στη συναλλαγή. Ε, και πολλές φορές δεν έχει κανείς την επιλογή του τρόπου πληρωμής. Εγώ είμαι πρόθυμη να συζητήσω ό,τι θέλετε και καινούργια μοντέλα κτλ. Αλλά οι πιστωτέ να δεσμευτούν ότι θα προτείνουν σε όλου του πελάτε ένα τρόπο πληρωμή και θα χρεώνουν ε, την υπηρεσία με τρόπο γνωστό ε, σε όλους τους καταναλωτές για να μπορεί ο καθένας να επιλέγει ε, τον τρόπο πληρωμής που θέλει ανάλογα με το πόσο κοστίζει. Ζήτω η διαφάνεια, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Χάρτσινγκ. Um, Την αντίδραση της Γενικής Διεθνής Ανταγωνισμού έχω να πω τρία πράγματα. Όσον αφορά τη χρέωση αυτή, πέρσι τον ε, Νοέμβριο το είχε υπερασπιστεί η Γενική Διεύθυνση ε, δηλαδή ότι καλό είναι να έχουμε άμεση χρεώσεις και όχι χρέωση ανά συναλλαγή. Στην ίδια ακρόαση είχε πει ξεκάθαρα, ε, είχαν πει ξεκάθαρα οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων πως εμείς δεν θα δίνουμε επιδοτήσεις. Και αυτό βεβαίω σκέφτονται και οι αρχέ του ανταγωνισμού. Δεύτερον, δεν άκουσα καμία δημόσια διοίκηση να χρησιμοποιεί το μέσο ότι δηλαδή σκοπεύουν να δώσουν εκπτώσεις στους καταναλωτές εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο. Δεύτερον, εκπλήσω με λίγο που ακούω πως ή ένα μοντέλο άμεσης χρέωσης που βασίζεται στο ΜΙΦ δεν είναι διαφανές. Η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών ήταν σαφής. Θα πρέπει να είναι maximum 8,8 ε, cents του ευρώ ανά συναλλαγή μετά την μετάβαση. Αυτό είναι και στο site. Οπότε νομίζω πως είναι διάφανο. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση στο τέλος. Το Κοινοβούλιο πρέπει να σκεφτεί το εξής. Είναι προς το συμφέρον των ε, καταναλωτών γιατί δεν είναι ε, ζήτημα των τραπεζών ε, από πλευράς του. Είναι λοιπόν προς το σημερινό των καταναλωτών μέρος του κόστους να καλύπτεται από ένα τέλος το οποίο πληρώνει η τράπεζα του πιστωτή που εξυπηρετεί την ε, δημόσια διοίκηση ή την επιχείρηση. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει. Ε, Μάλιστα. Κύριε Χάρτσεν, σε εμπιστευόμαστε. Και εμεί θα μα εμπιστεύεστε ότι είμαστε υπέρ των καταναλωτών και προ όφελό του, γιατί και όλοι εμεί καταναλωτέ είμαστε. Να είστε βέβαιος. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μεβίλ, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέει, το Συμβούλιο είναι καλύτερο από εσά, τι σα είπανε. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση που μόλις ακούσαμε δείχνει πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Ακούσαμε εκπροσώπους των χρηστών, της βιομηχανίας, του κλάδου δηλαδή των τραπεζών που μιλούν Ακούσαμε εκπροσώπους των τραπεζών να μιλούν εξ ονόματος των καταναλωτών, που καμιά φορά είναι και παράδοξο, και εκπροσώπους ε, που μίλησαν για συμφέροντα καταναλωτών διαφορετικά από αυτά που ανέφεραν κάποιοι προλαλήσαντες πριν από 10 λεπτά. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να βγάλει κανείς συμπεράσματα από αυτά που ακούμε και από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Πάντως, είναι σαφές ότι υπάρχει συνένεση και αυτό είναι πολύ ευθαρρυντικό για την ανάγκη ε, ε, καταληκτικής ημερομηνία για να μεταφερθούμε στο σύστημα ΣΕΠ. Αυτό δεν το αμφισβήτησε κανείς εντός ηθούσης, ότι χρειάζεται επίσης να ρυθμιστεί αυτό. Τώρα, ο τρόπος που θα γίνει επιδέχεται και ρύθμιση και ερμηνείε, αλλά ότι είναι απαραίτητοι οι κανόνες και μια καταληκτική ημερομηνία φιλόδοξη, νομίζω είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα, αν θα πρέπει να έχουμε μία ή δύο ημερομηνίε, ρωτήθηκε. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Ο βασικός στόχος της πρότασης κανονισμού είναι η ημερομηνία. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσαμε ότι δεδομένου ότι το προϊόν του εμβάσματος είναι ένα στάδιο πιο πέρα υπάρχει μια μετάβαση πιο γρήγορη. Λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε αυτή την ορμή που έχουμε τώρα, αυτή τη φόρα που έχουμε πάρει, για να βάλουμε μια ημερομηνία φιλόδοξη, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες και ιδιαίτερα ε, οι δημόσιες διοικήσεις, οι κρατικές μηχανές να κάνουν ε, ε, μια προσπάθεια για να μεταβούν στο νέο σύστημα γρήγορα και αυτό θα συμπαρασύρει εκτός από τα εμβάσματα και το άλλο προϊόν που είναι οι πάγιες εντολές. Ε, για τα εμβάσματα θα μπορούσαμε να πούμε ένα χρόνο μετά την έγκριση του κανονισμού και αυτό θα δημιουργούσε και μια επιπλέον δυναμική υπέρ της ΕΠΑ και θα ενθάρρυνε όλους τους χρήστες ε, αλλά και τους παρόχους ε, της υπηρεσίας να επιταχύνουν και το άλλο σκέλος που είναι η μετάβαση στο σύστημα και για τις πάγιες εντολές πληρωμών. Ένα συμπληρωματικό μέτρο που ανέφερε η κυρία Ισαΐα, δεν απατώμε, είναι το θέμα της ενημέρωσης. Είναι σαφές, αν θέλουμε να έχουμε μια μετάβαση αναγκαστική ή εθελουσία, σε κάποια κράτη-μέλη χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνουν προσπάθειες για ενημέρωση. Η ανάλυση που έχουμε κάνει για την κατάσταση της μετάφασης στο σύστημα ΣΕΠΑ, τι λέει. Ε, αυτή έχει επιταχυνθεί σε χώρες όπου είχαν γίνει προσπάθειες ουσιαστικές όμως ενημέρωσης και πληροφόρηση και από τις τράπεζες αλλά και από τις εταιρείες, επιχειρήσεις. Και μάλιστα τα κράτη-μέλη εκείνα που όλοι οι χρήστες συμμετείχαν στην εφαρμογή του συστήματος ΣΕΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Και εκείνα τα κράτη-μέλη που υπολείπονται είναι χώρες όπου δεν υπάρχει πληροφόρηση και όπου οι χρήστες είναι αποκλεισμένοι, είναι εκτός των διαφόρων ε, συμβουλίων μετάβασης προς το ΣΕΠΑ. Πολλά τεχνικά αναφέρθηκαν, δεν θέλω εγώ να επεκταθώ σε αυτά. Ένα μόνο σημείο για το ρόλο του Συμβουλίου ΣΕΠΑ, το οποίο Συμβούλιο συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Συμβούλιο ΣΕΠΑ είναι προσανατολισμού όργανο στρατηγικό ε, και απαρτίζεται από εκπροσώπους πολύ υψηλού επίπεδου ε, των ε, τραπεζών. Συμμετέχουν και καταναλωτές και επιχειρήσεις και έμποροι και εκπρόσωποι του δημοσίου και όλοι οι χρήστες δεν νομίζω ότι έχει ρόλο εκεί ε, στην ενημέρωση ε, προδιαγραφών τόσο τεχνικής φύσεως. Καλή η διαβούλευση, αλλά δεν είναι ο ρόλος του αυτός. Δεν είχαμε υπόψη μας όταν συστήσαμε αυτό το όργανο να του δώσουμε ρόλο τεχνικής τυποποίησης. Δεν είναι εκεί οι κατάλληλοι εμπειρογνώμονε σε αυτό το Συμβούλιο για να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις ή να συμβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον κλάδο για την ε, ενημέρωση κάποιων τεχνικών προτύπων ή τη θέσπιση κάποιων τεχνικών προτύπων. Η κατεξουσιοδότηση πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, στην πρόταση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάτι, τέτοιες προτάσεις για την ενημέρωση τεχνικών προδιαγραφών, μη ουσιαστικών όμως που αναγράφονται στο παράρτημα, είναι πρόθυμη απολύτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξτάσει ποια είναι ουσιώδη και ποια επουσιώδη ή λιγότερο σημαντικά, αλλά σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να ανατίθενται αυτές τις εξουσίες κατά εξουσιοδότηση σε άλλους με δικαίωμα ανάκληση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για ε, την άσκηση αυτών των εξουσιών. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει κάποια ευελιξία για να μπορέσει ο κλάδος να ε, ξεχρονίσει τους κανόνες που ισχύουν και ε, μπορεί να χρειάζεται και τροποποίηση του παραρτήματος στον κανονισμό. Επίσης, είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι ο κανονισμός εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους κανόνες ε, που ίσχυσαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών ε, για τα εμβάσματα και για τις πάγιες εντολές πληρωμής. Επίσης, ε, προσθέσαμε και περιορισμένες διατάξεις για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα νέα προϊόντα γιατί σήμερα η πάγια εντολή ακόμα δεν είναι δυνατή διασυνοριακά, οπότε για κάποιες περιορισμένες διατάξεις χρειάζεται μάλλον να ε, προβλέψουμε ασφαλιστικές ε, ρήτρε και ασφαλιστικές δικλείδες για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτά τα νέα προϊόντα. Δεν θα επανέλθω στο θέμα των τελών και των συναλλαγών. Ε, θα ήθελα μόνο να διορθώσω κάτι που υπόθηκε. Σε 70% των ε, συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, τέτοιου είδους χρέωση. Όχι, είναι 30%, δεν είναι 70%. Το υπόλοιπο 40% είναι κατάσταση στη Γερμανία και στη Γερμανία δεν είναι η ίδια κατάσταση. Δεν χρεώνουν τις συναλλαγές, χρεώνουν τις συναλλαγές που απορρίπτονται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε, κυρία Πρόεδρε, όταν θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση τη κυρία Εσαία. Πάντω, γενικά βλέπω ότι είναι ευρία η συνένεση να... για... την ανάγκη ακριβώς να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα με ε, ημερομηνία για τη μετάβαση φιλόδοξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ δεδομένες της ε, της περιπλοκότητας ε, του θέματος ε, σίγουρα αυτή εδώ η ακρόαση ήταν πολύ χρήσιμη ενδιαφέρουσα και θα επιτρέψει στην εισηγήτρια να προετοιμάσει σωστά το θέμα για τις δικές μας συζητήσεις. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, όλους τους εμπειρογνώμενους που ήρθαν και θα περάσουμε αμέσως Ευχαριστώ. Αντίο σα Και θα περάσουμε αμέσω στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Ο κύριο ε, Σάντζες Πρεζέντο. Αν μπορείτε να Αποχωρήστε ησύχως, θα μας κάνετε πολύ μεγάλη χάρη. Euh, voilà, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est possible de sortir sans Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να φύγετε χωρίς να συζητάτε. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί εμείς έχουμε συνεδρίες. Il Euh, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δίνω το λόγο στον εισηγητή και έχουμε και τέσσερις σκιώδεις εισηγητές παρόντες, οπότε μπορούμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρώτη τοποθέτηση είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Τρία είναι τα μεγάλα θέματα. Πρώτο, είναι οι προπαρασκευαστικές δράσεις και εργασίες που έχουν αρχίσει από τότε που ε, διορίστηκε ο εισηγητής για το δανεισμό μετά θα μιλήσω για ένα άλλο στοιχείο προκατακτικό επίσης που είναι το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας. Και το τρίτο θα είναι, κατά την άποψή μου, θα σας πω ποιοι είναι οι προσανατολισμοί που πρέπει να έχει αυτή η πρωτοβουλία η ρυθμιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλους για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε ε, τους σκιώδης ηγητές, τη γραμματεία, τους ε, βοηθούς μας. Συνεδριάσαμε με τους σκιώδης ηγητές για μία πρώτη διερευνητική συζήτηση. Κάναμε και σεμινάριο στις 26 Ιανουαρίου ε, για την ε, υπεύθυνη πίστη ε, και το Δεκέμβριο είχαμε συναντήσεις και τον Ιανουάριο με τον κύριο Μπαρνιέ. Συζητήσαμε σε βάθος αυτά τα θέματα που σήμερα μας απασχολούν. Μπορώ να σας πω ότι είχα μέχρι και 24 συνεδριάσεις με τους ενδιαφερομένους. Έχω όλα τα στοιχεία ε, των ενδιαφερομένων στη διάθεσή σας ε, ε, πολύ μεγάλη προεργασία λοιπόν και η ενημέρωση. Προετοιμάζουμε το χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση. Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο έκθεσης ε, έχει προχωρήσει στην προετοιμασία του. Στη γραμματεία ανατέθηκε μια μελέτη για τον ανταγωνισμό και ελπίζω εν ευθέτω χρόνο να έχουν όλοι οι βουλευτές την έκθεση αυτή στη διάθεσή τους για να ετοιμάσουν τις τροπολογίες τους και ε, πραγματικά θέλω να είναι πολύ φιλόδοξη η κοινοβουλευτική διάσταση εδώ. Διαπιστώνεται ότι εγώ ορίστηκα εισηγητής για ένα θέμα που ονομαζόταν ε, μέτρα για το υπεύθυνο δανείζει και δανείζεστε, lending and borrowing. Τώρα γίνεται λόγο μόνο για την πίστη που έχει να κάνει με ακίνητα για κατοικία. Δεν καταλαβαίνω. Δεν συμπίπτει ακριβώς το θέμα το ένα με το άλλο. Βεβαίως θα πρέπει ε, να είναι ε, υπεύθυνη η στάση και των δανειοδοτών και των ε, δανειοληπτών. Είδαμε τι έγινε με τις υποθήκες, τα subprimes και τα παράγωγα και έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή το ενυπόθηκο δάνειο. Αλλά ε, ήταν πολύ περισσότερο από κρίση των υπόθηκου δανείου αυτή η κρίση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009 μια μελέτη έλεγε ότι μεταξύ των χαρακτηριστικών που οδήγησαν στην κρίση δύο συνδέονται πολύ με το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, η διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και ε, στα majors και επίσης ε, η συνολική ε, υπερχρέωση του συστήματος σε όλες τις χορηγήσεις, όχι μόνο στα ενυπόθηκα δάνεια. Φούσκωσε πάρα πολύ δηλαδή το σύστημα. Ε, στην Επιτροπή Κρίσης αυτή τη βδομάδα είδαμε και μάθαμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ηνωμένες Πολιτείες που είχε αναλάβει να εκπονήσει μια έκθεση για την κρίση είχε υποβάλει τα συμπεράσματα και είπε ότι η υπερχρέωση, η υπερβολική χρέωση όρων ευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό για την κρίση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα ενυπόθηκα δάνεια, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή, ή τα στεγαστικά θέλετε. Ε, συζητούμε για την οικονομική διακυβέρνηση, αυτό το πακέτο νομοθετημάτων και συμμετέχει εκεί και το ιδιωτικό χρέος για να δούμε πώς έχει ε, εξελιχθεί ε, το ιδιωτικό χρέος στα πλαίσια του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη που ξέρουμε πόσο υψηλό είναι και από την άλλη όταν μιλάμε για οικονομική ισορροπία να λαμβάνουμε υπόψη και κριτήριο και το ιδιωτικό χρέος, όχι μόνο το κρατικό. Ε, είναι λοιπόν ένας παράγον που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σε αντίθεση με το δημόσιο χρέο, όπου έχουμε δείκτε, έχουμε ένα σύστημα που δείχνει ποια είναι τα όρια ή ποια είναι τα ορόσημα για τα δημόσια χρέη, στο ιδιωτικό χρέος αυτό δεν ε, ε, υπάρχει. Και εμείς έχουμε μια οικονομία υφόρο και βιώσιμη. Τον Οκτώβριο του 2010 εγκρίναμε την πρώτη έκθεση της Επιτροπής Κρίσης μέσω πρόθεσμη που έλεγε ότι ένα από τα σοβαρά αποτελέσματα της κρίσης, όχι μόνο αιτία, ήταν η μεγαλύτερη χρέωση. Δηλαδή, η χρέος δεν σημαίνει μόνο να αυξάνει τα επισφαλή δάνεια, στεγαστικά δάνεια, ε, αλλά και άλλα δάνεια καταναλωτικά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα της χώρας που γνωρίζω περισσότερο, στην Ισπανία. Το default, δηλαδή η αδυναμία ε, πληρωμών, είναι 2,5%. Ενώ 5% ε, το διπλάσιο είναι στα δάνεια τα στεγαστικά και τα στεγαστικά ε, δάνεια στους επιχειρηματίες, στους εργολάβους ε, ε, το, η αδυναμία πληρωμών, η επισφάλεια είναι στο 10%. Δηλαδή, τα βασικά προβλήματα δεν είναι στον μεμονωμένο πολίτη που παίρνει ένα στεγαστικό δάνειο, αλλά είναι και ευρύτερα τα θέματα και καλύπτονται από τη σημερινή νομοθετική δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ήδη από το 2001 η Επιτροπή Βασιλείας είχε κάνει μια έκθεση σχετική ε, για πολύ χρεωμένα ιδρύματα και οργανισμούς και στις Ηνωμένες μάλλον συγγνώμη, στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν αντίστοιχες προσπάθειες. Ε, δεν μιλάμε εμείς για το δημόσιο χρέος όμως. Ε, για το ιδιωτικό χρέος. Και πρέπει να σας πω ότι μια πρωτοβουλία που θέλει να καλύψει την υπερχρέωση δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με τα στεγοστικά δάνεια των ε, μεμονωμένων πολιτών. Ε, αυτό θα ήταν ατελές. Στις 23 λοιπόν Νοεμβρίου του 2010 και σε συνεργασία με τους σκιώδεις ηγητές έστειλα μια επιστολή στον κύριο Μπαρνιέ λέγοντας ότι θα πρέπει να διευρυνθεί ε, όχι μόνο το retail, τα ιταλιανικά ενυπόθηκα ή στεγαστικά δάνεια. Μας απάντησε ο κύριος Μπαρνιά, είχαμε και συναντήσεις μαζί του και κατέθεσε μια πρωτοβουλία. Και ανέκαθεν του λέγαμε του κυρίου Μπαρνιέ ότι μια πρωτοβουλία τέτοια για τα στεγαστικά δάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι μόνο το retail, δεν είναι μόνο σε επίπεδο μικρού καταναλωτή, είναι το ε, πρώτο βήμα μόνο. Και μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στείλαμε στον κύριο Μπαρνιέ ε, μια επιστολή, δηλαδή και στον κύριο Μπαρνιέ και στον κύριο Μπαρόσο, το γνωρίζουν οι σκιώδεις γιατί πήραν και εκείνη την ίδια επιστολή, ότι να είναι το πρώτο βήμα μόνο και να δούμε ποιες ήταν αυτές οι στρεβλές πρακτικές χορήγησης δανείων και να βεβαιωθούμε αυτές οι πρακτικές να μην επιζημίε ε, επιζημίες ούτε για τους ε, φορολογουμένους ούτε για τους ε, Ε, καταναλωτές ή τους πολίτες που έχουν ε, οικονομίες και αποταμίευσεις στις τράπεζες. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πρώτον δεν καλύπτει όλο το πεδίο ευθύνης που θα έπρεπε για να δούμε τα προβλήματα που συνδέονται με το ζήτημα ε, της υπεύθυνης χορήγησης δανείων, δανειοδότησης και δανειοληψίας. Επίσης, αυτό το θέμα των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη 68% των πολιτών έχουν ιδιόκτητη κατοικία που την έχουν πάρει με στεγαστικό δάνειο, με υποθήκη. 50% είναι οι υποθήκες του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Και 12.000 ευρώ κατά κεφαλή χρέος, οι υποθήκες σημαίνουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, αυτό το κανονισμό που μας ε, προτείνουν. Εγώ θα είχα τρεις αρχές να προτείνω και να σας δώσω πέντε μεγάλους προσανατολισμούς. Οι τρεις αρχές έχουν ως εξή. Πρώτον, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται ενιαία τα προϊόντα. Αυτό που μας ενδιαφέρει και είναι ισχύ του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας και της καινοτομίας. Δεν υπάρχει ένα και μόνο μοντέλο για να λυθούν όλα τα προβλήματα ενιαίο. Οπότε ο δικός μας προσανατολισμός δεν θα πρέπει να επιζητεί την ομοιομορφία των προϊόντων. Δεύτερον, δεύτερη αρχή. Δεν θέλουμε επίσης ο κανονισμός να αλλοιώσει ε, τις αρχές ή τα νομικά καθεστώτα που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θα διασαλεύσει την ένομη τάξη ο κανονισμός. Τα προβλήματα είναι γνωστά και τα συστήματα είναι απαντήσεις ετών. Δηλαδή, επειδή μπορεί να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να ανατρέψουμε την τάξη των κρατών, να βρούμε ποια είναι τα προβλήματα, να τα λύσουμε και να μην δημιουργούμε, να μην προκαλούμε νέα και ανεπιθύμητα στην ένωμη τάξη των κρατών μελών. Οπότε σεβασμό στις παραδόσεις, στις αρχές, στις νομικές ε, της κάθε χώρας. Και αυτό θα ήταν η δεύτερη αρχή. Τρίτη αρχή. Θα πρέπει να ορίσουμε σαφώς πώς θέλουμε να κινηθούμε. Ο κανονισμός αυτός δεν θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα συνέχεια. Τι είχα, Γιάννη, τι είχα πάντα, business as usual. Θα πρέπει να αλλάξουμε το κοινοτικό κεκτημένο για τις πιστώσεις. Όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα χρειάζονται απάντηση ε, προοδευτική χωρίς να ανατραπούν βέβαια όλα τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή να μην γκρεμιστεί το κοινοτικό κεκτημένο αλλά να θεωρηθούν τα όσα ισχύουν για τα δάνεια. Ωραία. Αφού τα είπα όλα αυτά, ποιοι είναι οι προσανατολισμοί τώρα. Πέντε σας είπα, κατά την άποψή μου. Με μεγάλη σαφήνεια θα σας ε, περιγράψω και ε, αν χρειαστεί θα σας εξηγήσω και τα θέματα, αφού σας ακούσω και σας ε, πού θα πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή αυτά τα πέντε ζητήματα και πού θα πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή μας. Πέντε προσανατολισμοί. Πρώτον, καλή είναι η πρόταση της Λευκής Βίβλου του 2007 για τις αγορές τις ανταγωνιστικές. Τη δεκαετία του 70 ε, τι θέλαμε στην εσωτερική αγορά. Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και ελεύθερη εγκατάσταση ε, με τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Στη δεκαετία του 80 η εσωτερική αγορά βασίστηκε κυρίως στο να λειτουργήσει μια ελάχιστη εναρμόνιση. Οπότε θέλαμε να αποφύγουμε μια λειτουργία πώς να το πω, ε, συγκρουσιακή της αγοράς, να λειτουργεί απρόσκοπτα και λογικά. Και από το ενιαίο νόμισμα και μετά, αυτό που θέλουμε είναι μια νέα ε, φάση το κεφάλαιο να επιτρέπει να βοηθάει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αλλά αυτό απαντά σε μια οικονομική λογική, αμυγός να δημιουργείται αξία μέσω της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας. Αυτή λοιπόν η λευκή βίβλος που ζητάει αύξηση ε, τη αποτελεσματικότητα στον ανταγωνισμό καλό είναι ως προσανατολισμός και θα προσπαθήσουμε πιστεύω εγώ να το ενισχύσουμε. Δεύτερος προσανατολισμός. Διάβασα με μεγάλη προσοχή την έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο που μελετούσε πώς πρέπει να ρυθμίσει το θέμα των στεγαστικών δανείων. Και έκανε τρεις προτάσεις και πάλι που νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τις υιοθετήσουμε και να τις υπερασπιστούμε. Έλεγε πρώτον ότι θα πρέπει οι οικονομίες ε, των καταναλωτών να προστατεύονται από την ε, άφρονα δανειοδότηση. Επίσης θα πρέπει να είναι δεδομένη η φερεγκιότητα των τραπεζών, να μην δίνουν αλόγιστα δάνεια επίσης. Και τρίτον να γίνει μια προσπάθεια να μειωθούν αυτά τα πικ ε, στην οικονομία, ε, να εξισορροπηθούν και με ένα τρόπο που να λειτουργεί καλύτερα η οικονομία, να μην έχουμε ε, απότομες αυξομοιώσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλαγές Προστασία λοιπόν και των αποταμιεύσεων των ε, καταναλωτών, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και της χρηματοοικονομίας βεβαίως, χωρίς όμως να είναι τόσο σε αυτές οι φούσκες όταν σκάνε και να συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Θα πρέπει σιγά σιγά να στέλνουμε και τέτοια μηνύματα ε, και φρένα για να ε, μην έχουμε επανάληψη τέτοιας ε, κρίσης με τη σφοδρότητα που τη γνωρίσαμε. Και το ίδιο που κάνουμε για το δημόσιο χρέος κανονικά θα πρέπει να γίνει και στο ιδιωτικό χρέος. Άλλο στοιχείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι από τη Λευκή Βίβλο ε, το πρώτο, ε, το δεύτερο είναι η έκθεση ε, Turner που σας είπα και το τρίτο είναι τα συμπεράσματα του G20. Γίνεται λόγος για βελτίωση της ρύθμισης και της εποπτείας, προφανώς, αλλά αυτό είναι γενικό λόγο. Κάτι πιο ειδικό είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα και μεγαλύτερη ευελιξία. Ευελιξία τι σημαίνει κατά την άποψή μου το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει πραγματικά να επιτρέπει να απαντάμε ε, στις ανάγκες των οικογενειών, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος θεμάτων να μπει εδώ αν θέλουμε πραγματικά να ε, υλοποιήσουμε αυτά που δεσμεύτηκε να κάνει το G20. Ένα τέταρτο σημείο που επίσης θα πρέπει να βάλουμε και δεν ε, συμπεριλαμβάνεται αρκετά και σε μερικές περιπτώσεις καθόλου. Γι' αυτό είναι η μεταρρύθμιση να συνάδει με τη νέα ε, διάταξη της σύνεσης και της εποπτείας στην Ευρώπη. Ωραία, βάλαμε ένα σύστημα ευρωπαϊκής εποπτείας, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να πούμε πώς θα δρά αυτό ε, για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν ε, με τα ε, άφρονα δάνεια και να δούμε τι θα κάνουν οι νέες αρχές που μπαίνουν στο σύστημα και πώς θα ενισχυθεί το ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο στην Ευρώπη. Είναι μια διαδικασία αυτή προοδευτική δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα και μετά να διαφωνήσουμε και να το ε, ξυλώσουμε. Δεν θα γίνουμε ε, πινελόποι, ας πούμε, που ότι, ότι ήφαινε την ημέρα το βράδυ το ξύλωνε. Όλα αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να δίνουν εμπιστοσύνη ε, στην αγορά των στεγαστικών δανείων στην Ευρώπη και θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτή η αγορά των ανυπόθηκων δανείων στην Ευρώπη είναι ε, ισχυρή, στιβαρή, αξιόπιστη, αξίζει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και των επενδυτών και να θεωρούν ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ευκαιρία. Και άρα θα πρέπει να ενισχυθεί και σε αυτό το τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν τα πέντε στοιχεία που ε, θεωρώ προσανατολισμούς. Και κλείνει το μικρόφωνο. Και στη συνέχεια, αν θέλετε, να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες αφού σας ακούσω. Για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους προσανατολισμούς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε συγητή. Ήσασταν πολύ αναλυτικός, αλλά έχουμε τέσσερις και τι συγητές παρόντες και θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 5.30 και θα ήθελα να τους δώσω το λόγο σε όλους. Οπότε... Πρώτα ο κύριος Αλφρέντο Παλώνε. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή την παρουσίαση του συναδέλφου ε, Σάντσες. Έχουμε ήδη συναντηθεί, έχουμε κάνει ήδη ανταλλαγές ε, απόψεων, έχουμε εξαιρετική συνεργασία και πιστεύω μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο για να φτάσουμε σε κοινό ψήφισμα. Να πω αμέσως ότι συμμερίζομαι μέγα τμήμα των... Ε, της επιστολής που μας έστειλε ο συνάδελφος Πρεζέντο μαζί με την Πρόεδρο Θεωρώ όμως ότι σε αυτή την επιστολή Υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα που λέει ότι η μεγαλύτερη αφαιρεγγιότητα οφείλεται σε δάνεια και σε επενδυτές που ζήτησαν ε, δάνεια για να κάνουν ε, κατασκευαστικές, ε, κατασκευαστικά έργα. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την πρόταση που έχει αναγγελθεί. Εδώ είναι το κλειδί, εδώ είναι η σύγκρουση για να κάνουμε κοινέ προτάσει. Με όλο το σεβασμό βεβαίως στην κρίση που διανύουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα αίτια ήταν ακριβώς η φούσκα των ακινήτων. Αλλά όπως λέει και αυτό το η επιστολή αυτή δεν προκλήθηκε από την αφαιρεγγιότητα των καταναλωτών. Κάθε άλλο. Μην ξεχνάμε πως το πρόγραμμα ξέσπασε στις ΗΠΑ και σε μας έφτασε ο αντίκτυπος εδώ στην Ευρώπη εντάξει, ο καταναλωτής να προστατευτεί και άρα να βρίσκεται σε μια θέση διαφάνειας για τις διαδικασίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Εδώ συμφωνώ όσον αφορά τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών. Προσοχή όμως, γιατί εμένα πολύ με ανησυχεί ένα θέμα. Σωστή η ρύθμιση, εντάξει. Αλλά είμαστε όμως στην ε, ελεύθερη αγορά και γι' αυτό και νομίζω πως ε, Φοβάμαι μάλλον μήπως τελικά έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν ε, προχωρήσουμε σε υπερβολικές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα γιατί η διαδικασία στην ουσία αφορά και εξαρτάται και από την ηθική του ανθρώπου και δεν μπορούμε δηλαδή να περιορίσουμε την ελευθερία των επιχειρήσεων και των τραπεζών η επιλογή για ένα δάνειο είναι σημαντική, αλλά είναι πολύ σημαντική για τον ίδιο τον καταναλωτή και πολύ συχνά είναι υποκειμενική. Και γι' αυτό και είναι σωστό να είναι ρυθμισμένη και θα πρέπει ο καταναλωτής, κάθε ένας δηλαδή ο οποίος ε, θα πάει να συνάψει ένα δάνειο, να είναι σε θέση, στην καλύτερη δυνατή θέση. Δηλαδή να έχει ο καταναλωτής όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Άρα λοιπόν νομίζω πως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένα κρίσιμα στοιχεία και δεν νομίζω πως είναι σκόπιμο να μπούμε σε αντίθεση ή σε σύγκρουση με, τους, ε, με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, με τους συναδέλφους δηλαδή. Απλώς να σας δώσω κάποιες ιδέες, γιατί εγώ έχω κάποια ανησυχίες όσον αφορά την προσυμβατική ενημέρωση. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα Όσον αφορά την εναρμόνιση, να επιβάλλουμε, λέτε, μια εναρμόνιση χώρα. Αν επιβληθεί από πλευρά τη Κομισιόν μια γενική εναρμόνιση, αφήνει μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Και αν όντω αφαιθούν τα κράτη-μέλη να κρίνουν μόνα του, τότε δεν υπάρχει μεγάλη εναρμόνιση. Μάλλον μπορεί να μην υπάρξει μεγάλη εναρμόνιση και είναι δύσκολη η επιτευχή του στόχου. Έπειτα μιλάτε σε κάποιο μέρος για κατάλληλες διευκρινήσεις. Για παράδειγμα, αγαπητέ Χάντσες, και εδώ πρέπει να πούμε το πρόβλημα της, ενημέρωση ενημέρωσης προ τη σύναψη του δανείου πρέπει να είναι προσωπική, προσωποποιημένη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει αυτό εκ των προτέρων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Και έπειτα, αξία του δανείου. Θα ήθελα εδώ να ζητήσω κάποια προβληματισμό από όλους τους συναδέλφους. Δηλαδή, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του ίδιου του δανειοδότη, όχι, αλλά και η σχέση ανάμεσα στην αξία του ακινήτου και του ποσού της, του δανείου. Για να προστατεύσουμε δηλαδή τις πιο αδύναμες ε, τάξεις της, κοινότητα, της κοινωνίας, για το θέμα των ενυπόθηκων δανείων, ιδιαίτερα εκείνων των νέων που έχουν ε, ευέλικτη εργασία, Υπάρχει και εγγύηση από τρίτα άτομα που μπορεί να είναι είτε οι γονεί ή συγκεκριμένα τρίτα άτομα. Το, το θέμα είναι να υπάρχει εγγύηση για αυτούς τους νέους. Έπειτα, η εξάλληψη του άρθρου 8 και δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για, με τεχνικούς όρους. Θα πρέπει να τα αφήσουμε στις κυβερνήσεις ή να εναρμονίσουμε αυτή την κατάσταση γιατί έχουμε και τραπεζικά συστήματα και από αυτόν δεν θέλω να ξεκινήσω οποιαδήποτε τσακόμο. Απλώς υπάρχουν οι δημόσιες και οι κρατικές μάλλον και οι ιδιωτικές τράπεζες με διαφορετική τελείως φιλοσοφία. Μια διαφορετική στάση λοιπόν για μια τράπεζα η οποία βασίζεται στην αποταμίευση και διαφορετική τελείως ε, για τις υπόλοιπε πιο εμπορικές τράπεζες. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα αναλύσουμε και να συζητήσουμε για αυτά τα προβλήματα. Πιστεύω ωστόσο ότι θα βρούμε κοινέ επιλογές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση για να ξέρουμε από πού προέρχεται ακριβώς η κρίση και η κρίση ακριβώς προξενήθηκε από αυτό το οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή ίσως σε κάποια να υπήρχαν προβλήματα με κάποια συγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια και το ότι το υποθηκευμένο ακίνητο πλέον κατέληξε να αξίζει λιγότερο από την αξία του δανείου. Βεβαίως, πολύ λιγότερο από το πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν γενικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει αυτό πως ε, δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να δούμε αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν και να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά για αυτά τα δάνεια. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μέλημά μας εδώ πέρα. Και μετά, όπως λέει και ο εισηγητής, το να αναλάβουμε άλλες πρωτοβουλίες και άλλες προτάσεις, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να δούμε μια άλλη στιγμή. υπάρχει νομίζω ούτως ή ε, υπάρχουν σχετικές οδηγίες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει νομίζω επικάλυψη. Λοιπόν πρέπει άρα να ακολουθήσουμε τις αρχές. Ευελιξία, να μην εμποδίζουμε δηλαδή καινοτομίε κτλ. Και, και δεύτερον διαφάνεια. Θα πρέπει δηλαδή και ο πίστοτης ε, και αυτός ο οποίος παίρνει το δάνειο να γνωρίζει πώς υπάρχει, υπάρχουν κάποιες απαιτήσει ποιότητας και θεωρώ πως υπαρχει υπαρχουν καποιες απαιτησει ποιοτητα είναι να έχουμε συγκρίσιμα συστήματα, δηλαδή συστήματα με βάση τα οποία να μπορεί να γίνει εύκολα η σύγκριση για το τι έχουν να προσφέρουν ε, διάφορες επιχειρήσεις, όχι μόνο δηλαδή η συνήθιση υποπτή, οι συνήθιες τράπεζες σε μια χώρα, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα μπορούν ε, να προσφέρουν ένα προϊόν το οποίο θα γνωρίζει και θα μπορεί να ευστηθεί ο καταναλωτής. Θεωρώ λοιπόν πως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ε, φερεγγιότητας αν θέλετε του κάθε δανείου αλλά βεβαίως το να είναι αυτό το μόνο κριτήριο σημαίνει πως υποτιμούμε και την εξειδικευμένη γνώση των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό τον τομέα δεν είναι αυτό το μόνο κριτήριο θα πρέπει να παραμείνουν οι πόρτες ανοιχτές για την εξειδίκευση των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα ε, με απαιτήσει ποιότητας και με διαφάνεια και θεωρώ επιπλέον πως θα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε κάποια ρύθμιση η οποία θα κάνει πάρα πολύ δύσκολη το να δίνονται δάνεια για να μην οδηγηθούμε δηλαδή σε μια πιστοτική στενοπό να μπορεί και ο κόσμος να πάρει ένα δάνεια γιατί όταν θέλει όταν θέλουν νέοι άνθρωποι να, να πάρουν ένα δάνειο να ε, έχουν την, ε, την δυνατότητα. Και στην περίπτωση βεβαίως ε, στην οποία κάποιο πιστοτικό ίδρυμα δεν θέλει να αναλάβει κανένα κίνδυνο ή δεν του επιτρέπουμε εμείς να αναλάβει κανένα κίνδυνο, δεν, δεν έχει κανένα ρόλο και καμία θέση στην αγορά. Δηλαδή ζωή χωρίς κίνδυνο και ο επιχειρήν χωρίς κίνδυνο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Ναι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε το ότι συζητάμε για τα στεγαστικά δάνεια. Έχουμε και μια άλλη οδηγία περί από την οποία είχαν εξαιρεθεί βεβαίως τα στεγαστικά δάνεια, αλλά αν δείτε την κρίση βλέπουμε πως ακριβώς αυτός ο τομέας απετέλεσε αιτία της ε, κρίσης. Ε, πρέπει λοιπόν να το δούμε. Από την άλλη βεβαίως πρέπει να είναι σαφές πως ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους στόχους και τους στόχους του κοινού συμφέροντος αλλά και τα ατομικά δικαιώματα. Δηλαδή πρέπει να λάβουν υπόψη τη σταθερότητα του συστήματος ε, γιατί αν δοθούν πάρα πολλές πιστώσεις ειδικά όταν υπάρχουν κειμενόμενα επιτόκια μπορούμε να οδηγηθούμε σε άσχημες επιπτώσεις και να οδηγηθούν ε, αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τα δάνεια σε κρίση. Αλλά από την άλλη πρέπει βεβαίως και ο κόσμος να έχει πρόσβαση στην πίστη να μην τη δυσκολεύσουμε υπερβολικά και ταυτόχρονα να προσφέρουμε ένα μάξιμουμ προστασία των καταναλωτών για να έχει ο κόσμος πρόσβαση σε καλά δάνεια και να μην παραπλανούνται. Οπότε στον τομέα της διαφήμισης θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες προδιαγραφές. Είναι θετικό αυτό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8. Επίσης ειδικά όσον αφορά κειμενόμενα επιτόκια θα πρέπει να έχουν ε, υπόψη τους οι χρήστες σενάρια και θετικά και αρνητικά ε, όσον αφορά την διακύμανση των επιτοκίων για να γνωρίζουν το τι θα τους τύχει εάν ανέβουν τα επιτόκια. Κάτι άλλο, οι προσυμβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης που αναφέρονται στο άρθρο 9 Νομίζω πως ε, είναι κάτι το θετικό αυτό το οποίο προτείνει εδώ πέρα η Κομισιόν. Πηγαίνουμε παραπέρα από αυτά τα οποία ρυθμίζονται μέχρι στιγμής και θα πρέπει να ενημερώνεται ε, ο πίστοτης και βεβαίως ε, το θέμα είναι πως όταν υπάρχουν κειμενόμενα επιτόκια να υπάρχει κάποια ενημέρωση όπως είπαμε για τα διάφορα σενάρια και επιπλέον θα πρέπει να έχουν δικαίωμα μιας δεσμευτικής προσφοράς αυτοί οι οποίοι ζητούν δάνειο για να μπορούν να συγκρίνουν διάφορες προσφορές, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι τόσο απλό και όταν μιλάμε για τον υπολογισμό του ετήσιου πραγματικού επιτοκίου θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια και σε βάθος χρόνου για την ε, διακύμανση αυτού του επιτοκίου έτσι ώστε σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει το άρθρο 12 υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση για το ποιο θα είναι τελικά το ποσό. Εμείς θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια επιτόκια τα οποία πρέπει να περιγράψουμε ως ε, κερδοσκοπικά και πρέπει να υπάρξουν κάποια όρια, ένα maximum όσον αφορά τα επιτόκια. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι μακροπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη σταθερότητα του συστήματος και άρα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, τις θέσουμε σε χειρότερη μοίρα από τις ε, βραχυπρόθεσμες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για μακροπρόθεσμες ε, σχέσεις ε, πίστης για να εμποδιστεί ακριβώς αυτό το boom, αυτή η άνθηση των βραχυπρόθεσμων δανείων. Και πρέπει να δούμε επίσης τι συμβαίνει όταν δίνονται δάνεια με βάση ε, μη επαρκή εξασφάλιση. Γιατί είδατε πως δίνονταν ε, δάνεια σε, με ύψος πάνω από το 100%, πάνω από το 100% του υποκείμενου της υποκείμενης αξίας. Οπότε οδηγούμαστε σε μια κατάσταση υπερχρέωσης. Εδώ πέρα πρέπει να ενισχυθούν ε, τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών για να μην ε, μένουν στο τέλος μόνοι τους όταν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και τέλος ένα ζήτημα ήταν βεβαίως ε, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, όπου ξαφνικά και απρόβλεπτα βλέπουν πως το πραγματικό κόστος στο, ίδιο, στο οικείο νόμισμα ξαφνικά αυξάνεται. Οπότε θα, υπάρχουν τουλάχιστον, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία πληροφόρηση για να μην χρεοκοπούν ε, οι πελάτες. Θεωρώ πως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για την οικονομική σταθερότητα και για τα ατομικά δικαιώματα των καταναλωτών. Χαίρομαι λοιπόν για την συνεργασία με τους ε, εισηγητές για την ε, σταθερότητα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Μάλιστα, τον λόγο έχει ο κύριος Χοντής και μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση για... Μετά από αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, γιατί θα ήθελα να τηρήσουμε την ώρα. Θέλω από την αρχή να πω ότι ο εισηγητής μας, τόσο με την εισήγηση την προφορική που μας έκανε σήμερα, όσο και με τη σοβαρή προσπάθεια συνεργασίας με τους κοιόδης εισηγητές και ακόμα με την πρωτοβουλία που ανέλαβε με το γράμμα που κατέθεσε προς τον κύριο Μπαρόζο ή έχω την εντύπωση και τον συγχαίρω ότι έχει αίσθηση του προβλήματος και στην έκταση και στο βάθος που απαιτείται πράγμα που δεν έχει η πρόταση που κάνει η Επιτροπή. Η πρόταση που καταθέτει η Επιτροπή είναι περιοριστική όσο αφορά το αντικείμενο αναφέρθηκε ο εισηγητής συμφωνώ με την επιστολή και δεύτερο κατά την άποψή μου τα προτινόμενα μέτρα είναι γενικόλογα επιφανειακά και εγώ νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε πιο τολμηρές κατευθύνσεις πιο αναλυτικά. Βεβαίως είναι απαραίτητος και αναγκαίος ο ρόλος των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά όταν καλύπτουν πάγιες κοινωνικές ανάγκες δεν μπορούμε να δεχτούμε να κινούνται με κερδοσκοπικό χαρακτήρα όπως αποδείχθηκε στην προκειμένη περίπτωση. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω για να κερδίζουμε χρόνο, όπως ανέφερε και ο εισηγητής και αναφέρουν σχετικές σοβαρές εκθέσεις και η έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και η έκθεση στη Μεγάλη Βρετανία είναι γιατί έχουμε έναν υπερδιωγκωμένο χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει αναπτύξει παιδεία που δεν τα είχε παλιά. Βασικές ανάγκες που δεν μπορεί πια να καλύψει λόγω της κατάρρευσής του το κοινωνικό κράτος, όπως το στεγαστικό δάνειο. Βασικές ανάγκες που δεν μπορεί να καλύψει ο καταναλωτής λόγω της συμπίεσης του εισοδήματο έρχεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας με κερδοσκοπικό τρόπο να πάει να τις καλύψει. Και τι γίνεται εδώ, επειδή η κερδοσκοπία, κάποιος συνάδελφος το είπε ρίσκο. Ναι, αλλά αυτό το ρίσκο για την αναζήτηση καινοτομίας και νέων προϊόντων ήταν η αιτία που είχαμε όλη αυτή την φούσκα και όλη αυτή την κρίση. Στην προκειμένη περίπτωση τι έγινε. Η καινοτομία έλεγε υπησέρχεται ο τραπεζικός τομέας στα ενυπόθηκα δάνεια, με αυτό δανείζονται οι ίδιες οι τράπεζες οι τράπεζες καταραίουν επειδή δεν μπορούν να εισπράξουν το ρευστό και έρχεται το κράτος να τα βοηθήσει. Επομένως, κατά τη δική μου άποψη, καλή η ρύθμιση, καλή η εποπτεία του τραπεζικού τομέα, αλλά μόνη της δεν φτάνει. Άρα πρέπει να κινηθούμε και προς άλλη κατεύθυνση. Μια τελευταία παρατήρηση, επειδή ξέρω ότι είναι ο σύντομο ο χρόνος, θα μας απασχολεί στη συνέχεια, αυτή την υπόθεση της θεσμικής κατοχύρωσης του Μεσίτη των δανείων δεν τη βλέπω και τόσο αθώα ή τουλάχιστον ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους για την εξέλιξη των πραγμάτων. Σταματώ εδώ γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια κίνηση κινητικότητα στην αίθουσα, αλλά επειδή βλέπω ότι και οι συνάδελφοι θέλουν να ψηφίσουν όπως είναι η ώρα η συγκεκριμένη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, είναι και η ώρα της ψηφοφορίας. Να πω ότι η 24η, 24η Μαΐου είναι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης, η κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 9 Ιουνίου, εξέταση των τροπολογιών στις 4 Ιουλίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 12 Ιουλίου και Ολομέλεια Οκτωβρίου προβλέπονται για την έκθεση αυτή. Oh, the seats nice and warm in the hot seats.

you your and Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία και όσοι φεύγουν ήρεμα παρακαλώ, όσοι μπαίνουν επίσης. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες και τον κατάλογο ψηφοφορίας. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Εάν είστε ευχαριστημένοι, παρακαλώ πατήστε το κουμπάκι. 33 members. 33 βουλευτές έχουμε μέχρι στιγμής, 36, 37, 37 και δεν βλέπω άλλες προσφορές. 39. Ανεβαίνει. 39 συνάδελφοι είναι παρόντες, 40, 36 μόνο πατάνε το κουμπί. Πατήστε το κουμπάκι παρακαλώ. Δεν έχει σημασία ποιο κουμπί. 39, ένας ακόμα. Εκτό μικροφώνου το σχόλιο. Α, λείπει ο Βέρνερ. Μάλιστα. Ε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. 33 είστε χαρούμενοι. Ένας είναι δυστυχής και πέντε δεν ξέρουν. Μάλιστα. Ξεκινάμε την έκθεση όλες Smith για συστήματα αποζημίωσης επενδυτών συμβιβαστική λύση F. Mm, mm. Παρακαλώ. Κυρία Περιβάνος. Ε, και ο θέλει πρώτα το λόγο. Όχι, Περβάνος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά στον κατάλογο ψηφοφορίας πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε οι τροπολογίες 77 6 ε, και 156 ε, να αποσυρθούν όπως το είχαμε ζητήσει στους σκιώδεις εισηγητές στην ε, τροπολογία του κυρίου Ζάλμπα για τις οποίες θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Μάλλον, και επίσης νομίζω πως επικρατεί κάποια υποκρισία για τον τρόπο με τον οποίο έχουν υποβληθεί αυτές οι τροπολογίες γιατί μετά από δικό μας αίτημα δεν αποσύρθηκαν αλλά υποβάλλονται με τρόπο αυτόνομο σε σχέση με τις ε, τροπολογίες του εισηγητή. Όταν όμως δει κανεί ε, την λογική του καταλόγου ψηφοφορία, τουλάχιστον οι τροπολογίες ε, του εισηγητή που είναι ταυτόσιμες θα έπρεπε να παρουσιάζονται πρώτες. Στις 48 ε, και 160 ή 13 και 63 οι τροπολογίες του εισηγητή είναι πρώτε. Ε, και οι τροπολογίες αυτές ε, δεν έχουν αποσυρθεί και τίθενται σε ψηφοφορία πριν από τις τροπολογίες του εισηγητή. Ζητώ λοιπόν από το ΕΛΚ να τις αποσύρει, τουλάχιστον να τις στρέψει τη σειρά της ψηφοφορίας ανάμεσα στις εισηγητέ, στις τροπολογίες του εισηγητή να ψηφιστούν πρώτα. Για τις τροπολογίες 76 και 156 μιλάω. Θα ακούσουμε τώρα τον εισηγητή. Εκτός αν θέλετε να ακούσετε πρώτα τον κύριο Μπάλτς. Μπέρκχατ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα αποσύρουμε τις τροπολογίες, κυρίως για τον εξής ε, λόγο. Γιατί πρόκειται για ταυτόσιμες τροπολογίες με άλλες άλλων ε, συναδέλφων. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για σκιαμαχία. Θα αφήσουμε λοιπόν τις τροπολογίες όσες έχουν. Όλε. Όλε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για το καλό τους έργο και νομίζω πως έχουμε καταλήξει σε καλές συμβιβαστικές λύσεις και βεβαίω αυτό οφείλεται στο ότι θεωρούμε πως θα πρέπει να τελειώσουμε στην πρώτη ανάγνωση και οι Ούγγροι παρουσίασαν όλους αυτούς τους φακέλους περί εγγύησης καταθέσεων κτλ. πριν ε, την διακοπή του καλοκαιριού. Οπότε σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας, τη Γραμματεία, την Κλέρ και τη γραμματεία του κόμματό μου των, των, των φιλελευθέρων. Υπάρχει και μια κλέρ στο γραφείο μου, πολλές κλέρ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι καταλήξαμε σε αυτές τις συμβαστικές ε, λύσεις. Η πρόταση της κυρίας Μπερές ε, έγινε και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε. Ε, νομίζω πλέον πως ε, θα κρίνει η Επιτροπή. Για εμένα είναι κάπως περίεργο γιατί η εν λόγω τροπολογία δεν, δεν είναι εδώ μέσα, έχει αναδιατυπωθεί σε άλλη. Και όσον αφορά αυτές τις δύο τροπολογίες είναι ταυτόσιμες με τις δικές μου. Κάποιο σχόλιο εκτός μικροφώνου κυρίας Μπερές. Μα, μα... Κυρία μου, δεν ε, ήμουν εγώ πρόεδρος εδώ μέσα, δυστυχώς. Και νομίζω πως ο κατάλογος ε, της ψηφοφορία δεν είναι δική μου απόφαση. Οπότε είπα, είμαι διατεθειμένος να σας ακούσω όλους και ειδικά α, την κυρία Πρόεδρο για το πώς θα κυλήσει ο κατάλογος ε, της ψηφοφορία. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ.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 Υπάρχουν, με συγχωρείτε, λίγοι λόγοι για να μην ε, ψηφίσουμε αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα. Ο κύριος Ολισμίτ έχει κάνει πάρα πολύ καλή εργασία. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω πως στους ε, συντονιστές είχαμε την ε, ευκαιρία να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, ούτως ή άλλως δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι συζητήσεις και νομίζω πω υπάρχει ανάγκη να τις ε, συνεχίσουμε. Σβέν, ναι, πρώτα απ' όλα σας να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον Όλε για τη συνεργασία που είχαμε. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις και οφείλω να πω πως ήταν κρίμα και σοκαριστήκαμε κάπως που είδαμε πως ε, πρώτα απ' όλα είχαμε μία συνάντηση με τον συνάδελφο Σάλμπα που ήταν ο αρμόδιος για το ΕΛΚ και μετά μάθαμε πως δεν ε, απέρριψε μία προσφορά για να καταθέσει τροπολογία έναντι χρημάτων, επιπληρωμή εδώ πέρα. Ε, δεν αποσύρθηκε αυτή, αλλά οφείλω να πω πως το βασικό πρόβλημα για εμένα δεν είναι το εάν θα ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία πρώτη ή κάποια άλλη. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε την ε, τροπολογία του όλε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το πραγματικό θέμα είναι πως σε ανάλογες περιπτώσεις δύο συνάδελφοι έχουν αποχωρήσει Κάποιο άλλος εκδιώχθηκε από τους σοσιαλιστές. Και ο κύριος Σάλμπα εξακολουθεί να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος παρά το ότι σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο είναι ήδη παραβίαση το, το να μην αρνηθεί κανείς τα χρήματα και μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο συνήθως ε, έχει ένα περιδικαίου αίσθημα και είναι περήφανο ε, γι' αυτό και θα έπρεπε νομίζω να κάνει τα δέοντα και σε αυτή την ε, περίπτωση. Οπότε το, το εάν θα ψηφίσουμε ή όχι δεν είναι το πραγματικό ε, ζήτημα εδώ μέσα. Υπάρχει ένας ε, σκιοσυγητής ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα πρέπει να γίνει τώρα πλήρη συζήτηση, λέει η πρόεδρο, για αυτό το θέμα, αλλά ο κύριο Μεντέστε Βίγκο ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω πω η παρέμβαση του κυρίου Κιγκούλτ είναι λαθασμένη. Νομίζω πως ε, έχει αναγνωριστεί πως ο κύριος Σάλβα δεν δέχτηκε χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει, έχουν στήσει παγίδες ε, στα διάφορα μέλη. Στη χώρα μου απαγορεύεται αυτό έτσι κι αλλιώς. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, οφείλω να πω πως συμφωνώ πως ε, τίποτα δεν φαίνεται να έχει αποδειχτεί και δεν πρέπει να προδικάζουμε ε, αυτό το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ε, από τις αρχές ε, και του Κοινοβουλίου και της Ισπανίας. Αλλά θέλω να πω πως διαβάζοντας τα όσα ακούστηκαν και εγώ είχα κάποια ερωτήματα για την ερμηνεία των όσων ελέγχθησαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο συνάλφος είπε πως θα ζητήσει βοήθεια είτε από την ομάδα του είτε από τις ισπανικές αρχές για το τι επιτρέπεται σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο. Οπότε δεν θα πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα αλλά να περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Θα πρέπει νομίζω να προχωρήσουμε με τον κατάλογο της ψηφοφορίας όπως έχει προετοιμαστεί. Όχι υπερβάνας, δεν σου δίνω το λόγο. Εκτός μικροφώνου κυρία Περές γιατί δεν περιμένετε μέχρι να τελειώσει η πρόεδρος, η πρόεδρος μιλάει και δεν θα λάβετε ξανά τον λόγο. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά που έχουμε, έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε κατά, κάποιες φορές περνάνε δεύτερες οι τροπολογίες του εισηγητή για να ψηφιστούν τροπολογίες άλλων. Αυτή είναι η διαδικασία, με βάση αυτό προετοιμαστήκαμε Εν μέρη σεβαστήκαμε τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας ψηφίζοντας, εάν το επιθυμείτε. Θα προχωρήσουμε τώρα με την ε, ψηφοφορία όπως την βλέπετε μπροστά σας. Περνάμε λοιπόν συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 60. Περβάς Μπερές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ένα της νομικής επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο της νομικής επιτροπής υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά να επαληθεύσουμε για να δούμε πως έχουν οι αριθμοί Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 καλύπτεται οπότε περνάμε στην 13 και 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτές 64 με προφορική τροπολογία του εισηγητή Ωραία, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρα η 66 καταπίπτει μάλιστα 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 66 καταπίπτει 3 της Νομικής Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 71 καλύπτεται από τη συμβαστική F. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε την 72. Ψήφισαν όλοι. Καταπίπτει. Ε, επειδή λείπει ο Βέρνερ συμβαίνουν αυτά. 16 και 73 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 74 καλύπτεται. 17 και 75 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 18 αποσύρεται 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή θα επαληθεύσω τροπολογία 76 δεκτή συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 της νομικής επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική D για να δω αν υπάρχουν προφορικές τροπολογίες σε όλες αυτές τις σελίδες. Ωραία, συμβαστική διπερ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ε στη σελίδα 16 την βρήκα εγώ. Την βρήκατε όλοι. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Γυρίστε τις σελίδες. Τροπολογία 35. Δεν την έχω βρει ακόμα. Σελίδα 22, τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10 της Νομικής Επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε τη 10 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. 150 καλύπτεται ήδη 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 11 της Νομικής Επιτροπής, της ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτή. 12 της Νομικής Επιτροπής υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 151 υπέρ, κατά αποχές 14 της Νομικής Επιτροπής Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. 152 και 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά α, συγγνώμη, ε, κατέψε 16 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές δεκτή 157 καλύπτεται 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 και 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 56 δεν την βλέπω, οπότε πάμε στην 57. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58 καλύπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 υπέρ. 5 αποχές. Κανένας κατά. Περιμένετε λίγο. Ψηφίζουμε και το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Να εξαφανίζεται κόσμος. Μπαίνουν, βγαίνουν κάρτες. Μάλιστα. 34 υπέρ 4 αποχές. Γιατί κάποιοι έφυγαν. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. That's it?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 Okay, excitement over. Ωραία, τελείωσε η αναστάτωση. Ρόμπερτ, αν είσαι έτοιμος, περνάμε στο σημείο 6. Ακεραιότητα και διαφάνεια της αγοράς της ενέργειας. Συγητής, ε, ο Ρόμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση κανονισμού όσον αφορά την ακαιρεότητα και τη διαφάνεια της αγοράς ενέργειας είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητη. Είναι προφανές ότι όταν, εκεί που υπάρχουν οι αγορές υπάρχουν πάντοτε και οι πειρασμοί να καταχραστεί κανείς την αγορά, να χρησιμοποιήσει ε, εσωτερικές πληροφορίες για να πλουτίσει. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας την οποία ε, η Κομισιόν μας παρουσίασε ως ένα απαραίτητο μέτρο που θα μείωνε το κόστος της ενέργειας και του φυσικού αερίου για τον καταναλωτή τελικά επέφερε το αντίθετο. Και συχνά είδαμε και λανθασμένες κινήσεις πάνω σε αυτή την αγορά που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τις πραγματικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό το, οι αγορές αυτές που πήραν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια να εποπτεύονται, να είναι διαφανεί και κάθε απόπειρα ε, ε, χειραγώγησης, κάθε κατάχρηση αγοράς να εντοπίζεται και να τιμωρείται. Ε, έτσι λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν είναι ευπρόσδεκτη, την υποστηρίζω σχεδόν στο σύνολό της. Ε, γνωρίζετε ότι η Επιτροπή μας απλά γνωμοδοτεί και η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας που μάλιστα έχει προχωρήσει πολύ στις συζητήσεις της. Είχαμε χτες ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για προτάσεις που κάνει ο εισηγητής Χατζημαρκάκης. Για την πρόταση αυτή κανονισμού, η Κομισιόν εμπνεύστηκε από την οδηγία για την κατάχρηση των αγορών και την χρήση εσωτερικών πληροφοριών που είχε προτείνει πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα ήμουν και εισηγητής την εποχή εκείνη. Ε, εμπνευστήκε λοιπόν από την ισχύουσα αυτή η οδηγία και στην πρότασή της άντλησε ε, και από την ε, μεταρρύθμιση της εν λόγω οδηγίας. Ξέρετε ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ σύντομα θα φροντίσει ώστε να ενισχυθεί η οδηγία αυτή. Και αυτό δημιουργεί ένα θεωρητικό πρόβλημα διότι η Κομισιόν Μπνεύστηκε από μια οδηγία που δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από τους συνομοθέτες και θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δεχτούν την πρόταση οδηγίας ε, συγγνώμη, του κανονισμού διορθώνει ο όπως παρουσιάζεται εδώ και να έχουμε μετά προβλήματα με την οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς. Αυτό βέβαια είναι για την ώρα θεωρητικό, θεωρητικός κίνδυνος, αλλά ήθελα παρόλα αυτά να τον ε, καταστήσω γνωστό συναδέλφος. Η πρόταση λοιπόν κανονισμού της Κομισιόν προτείνει η... να δημιουργηθεί ο Οργανισμός Ρυθμιστών για την Αγορά της Ενέργειας, την ΆΣΕΡ για να υποπτεύει την αγορά. Εγώ πιστεύω πως είναι λογικό κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η Άσερ, ο Άσερ, που θα ξεκινήσει αυτές τις δραστηριότητες με έδρα την Λουμπλιάνα, να έχει τα απαραίτητα μέσα και το απαραίτητο προσωπικό για να προβεί στην εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει βέλτιστη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στου εθνικούς οργανισμούς και την ΆΣΕΡ. αλλά και με τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ορθή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και την Ευρωπαϊκή Σχετική ε, Υπηρεσία ε, Οργανισμό, την ΕΣΜΑ. Στη συνέχεια θα πρέπει να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι χειραγωγούν την αγορά ή καταχρώνται θέσεις που έχουν. Και στη σύντομη αιτολόγησή μου διαπιστώνω ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στα μίνιμουμ και μέγιστα επίπεδα χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες. Και νομίζω ότι ακόμα κι αν θέλαμε να σεβαστούμε την εξουσία των κρατών να ορίζουν δηλαδή αυτά τις ποινές, γιατί αυτό θα παραμείνει μέσα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, θα πρέπει ωστόσο να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει ισότιμο πεδίο για τα θέματα ποινών. Κυρία Πρόεδρε, εγώ περιορίστηκα σε αυτά στις ε, τροπολογίες μου δεν θέλησα να μπω στη συζήτηση του κατά πόσο είναι απαραίτητο ή όχι να συμπεριληφθεί σε αυτό τον κανονισμό και η αγορά που σχετίζεται με τον ε, διοξιδιο του άνθρακα. Ε, αυτό που θέλει να κάνει ο συνάδελφος Χατζημαρκάκης, εγώ προσωπικά τον υποστηρίζω, τουλάχιστον στην επιλογή στο ότι δηλαδή είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί η αγορά του διοξίδιου του άνθρακα, γιατί είδαμε πρόσφατα πως, υπήρξαν, ε, πως έγινε μια κυβερνοεπίθεση ε, κατά αυτής της αγοράς, έγινε πολύ μεγάλη χειραγώγηση και πολύ μεγάλες απάτες ε, σε αυτή την αγορά. Και η Κομισιόν θα μας πει αν μπορεί να δεχτεί την προσέγγιση του Χατζημαρκά και αν θα επιθυμεί να φτιάξει χωριστή νομοθεσία για το διοξείδιο του άνθρακα. Εμένα προσωπικά θα με... εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να ρυθμιστεί και αυτή η αγορά. Τώρα, οι προτάσεις που εγώ πρότεινα, οι τροποποίησεις συγγνώμη, που πρότεινα στην πρόταση κανονισμού, στόχο έχουν να ορίσουν σαφώς ότι όλες οι συναλλαγές που γίνονται είτε είναι στο αγορά, στις πλευρές ε, πλατφόρμες διαπραγματεύσεων αλλά και οι συμφωνίες ε, και μεταξύ κυρίων που συνήθως είναι οι συμφωνίες που γίνονται σε αυτό το τομέα να είναι διαφανείς. Η Κομισιόν έχει κάνει προτάσεις Βέβαια, πριν να γίνει η πρόταση για κατεξοδότηση ε, πράξης, ε, θα πρέπει να γίνει μία διαβούλευση με τον ε, τομέα αυτό της ενέργειας, αλλά και με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εθνικές διαρχές θα υποχρεούνται να μεταγράψουν αυτόν τον κανονισμό στα κράτη-μέλη. Πρέπει και πάλι δηλαδή να μεριμνήσουμε ώστε να μην δημιουργηθεί μια ε, γεωγραφία του κακού μαθητή στην Ευρώπη, θα πρέπει όλα τα κράτη να εφαρμόσουν με τον ίδιο τρόπο την ίδια νομοθεσία και θα πρέπει να ισχύει για όλες τις αγορές ενέργειας, για μάλλον για την αγορά ενέργειας, είτε προέρχεται από την Ευρώπη είτε είναι από τρίτες χώρε. Προτείνω επίσης να τελειοποιηθεί κάπως η πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά ορισμένες δυνατές παραβιάσεις, παραβάσεις μάλλον, γιατί υπάρχουν κάποιες πρακτικές στην αγορά που συνίστανται τον Μένουν διάφορες ε, συναλλαγές μεταφορών ενέργειας που κάνουν ορισμένοι ε, πράκτορες ενώ τα αποθέματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Ε, κρατάνε δηλαδή στην άκρη κάποια αποθέματα. Και κατά τη γνώμη μου είναι και αυτό κατάχρηση της αγοράς. Α, ε, κάτι ακόμα που είναι προφανής κατάχρηση αγοράς είναι να υποφελείται κανείς ε, από γνώσεις ε, για μείωση δυνατοτήτων μετά από ατυχήματα ή δραστηριότητες συντήρησης. Το περασμένο Ιανουάριο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πολλαπλασιάστηκε μέσα σε κάποιες ώρες ε, επί 4. Από τα 15 έφτασε στα 60 ευρώ. Και την επαύριο μάθαμε ότι σημαντικές παραγωγικές μονάδες ε, ηλεκτρικής ε, ενέργειας είχαν σταματήσει να λειτουργούν και αυτό φυσικά ωφέλησε όσους γνώριζαν εκ των προτέρων αυτή τη βασική πληροφορία. Πιστεύω επίση πως είναι σημαντικό η Κομισιόν να λάβει υπόψη τις μελλοντικέ ε, εξελίξεις ε, τη ε, της αγοράς, της χονδρικής αγοράς καθώς και τις συνέπειες τη αγορά αυτής στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μάλλον ναι, στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να φροντίσουμε για τις κατεξοδόσεις της υπράξης σε αυτόν τον τομέα. Παίρνω σύντομα τις υπόλοιπε τροπολογίες που δεν είναι τόσο σημαντικές. Θέλω να πιστήσω μόνο την προσοχή σας στην τροπολογία που ζητώ από την Κομισιόν να θεσπίσει έναν μήνυμης όριο για να εξαιρούνται οι, από την παροχή δεδομένων οι φορείς οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεάσουν την αγορά της ενέργειας. Ως Κομισιόν είναι σε θέση νομίζω να ορίσει ένα τέτοιο κατόφλι και πιστεύω πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός de ορίου. Τελευταία σειρά τροπολογιών είναι αυτή που αφορά τις ποινές που ισχύουν για την ε, παράβαση των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού. Και εδώ προτείνω μια τροπολογία που έχω βρει ε, στην οδηγία που συζητάμε για το short selling όπου είπαμε ότι κυρώσει θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα τη παράβαση και να ξεπερνούν σημαντικά το πραγματικό ή δυνητικό όφελος κέρδος των παράνομων δραστηριοτήτων. Και έπειτα μια τελευταία τροπολογία που είναι κατά γνώμη μου σημαντική, ότι δηλαδή το προσωπικό και υπόρρητη οργανισμού προτείνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2015 να αξιολογήσει εκ νέου τις ανάγκες του σε πόρους και προσωπικό ώστε ενδεχομένως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν να προσαρμόσουν τους εν λόγω πόρους με βάση τις ανάγκες. και μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας για το 2012. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων και των σκιωδών για να προετοιμάσω μαζί τους μια ψηφοφορία που νομίζω ε, ότι θα είναι αρκετά εύκολη γιατί οι συζητήσεις στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας απέδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση ανάμεσα στις πολιτικές ε, ομάδες όσον αφορά την απαραίτητο χαρακτήρα αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη ιστοριούλα, μετά κάποια γενικά σχόλια και μετά κάποια πιο συγκεκριμένα για τις τροπολογίες. Η ιστορία είναι εξή. Είχα πρόσφατα μία συνομιλία με μία από τις μεγάλες εταιρείες ε, φυσικού αερίου στην Ευρώπη που εξέφρασε ανησυχίες για την ομοθεσία αυτή και η ανησυχία εκφράστηκε ως εξής. Μα Θεέ μου, εάν μία από τις ε, πλατφόρμες μας βγει εκτός προγραμματισμένα, εμείς το ξέρουμε και αγοράζουμε ε, το φυσικό αέριο από την αγορά σποτ. Εάν το μάθουν οι έμποροι θα αυξήσουν την τιμή και θα πληρώσουμε παραπάνω δεν θα μπορέσουμε να φυλάξουμε, να διφυλάξουμε τα συμφέροντά μας. Βεβαίως το αντίστροφο επιχείρημα είναι ποιος θα μας πει ότι η εταιρεία η οποία το γνωρίζει αυτό θα αγοράσει 120 μονάδες αντί για 100 ε, που χρειάζεται και θα πουλήσει τις 20 και θα βγάλει ένα ωραιότατο κέρδος. Οπότε εκεί πέρα μιλάμε πράγματι για εσωτερική πληροφόρηση. Πράγματι χρειάζεται αυτή η νομοθεσία, συμφωνώ με τον εισηγητή και πρέπει να συγχαρώ την Κομισιόν. Τρία γενικά σχόλια. Θεωρώ πως θα πρέπει να σκεφτούμε πως ο στόχος ε, τέτοιας νομοθεσίας και πρέπει να το πούμε ανοιχτά ε, είναι να προωθήσει τον ανταγωνισμό στις χοντρικές αγορές προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Γιατί για να γίνουν λιγότερο εφικτές οι συμφωνίες με εσωτερική πληροφόρηση και να είναι οι τιμές όσο δυνατόν πιο σταθερές ε, προς όφελος των καταναλωτών στην Ευρώπη. Δεύτερον, θεωρώ και θεωρώ πως υπάρχει κάποιο πεδίο εντός κανονισμού, αλλά το συζητάμε αυτό, πως πρέπει να σκεφτούμε την εναρμόνιση των προστήμων στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μην μπορεί μια αριθμιστική αρχή να έχει τις χει συνθήκες και αλλού να ισχύουν άλλες. Πρέπει να σκεφτούμε μια ενιαία προσέγγιση. Και τρίτη παρατήρηση. Εξυπονοείται νομίζω, αλλά πρέπει να το πούμε και ρητός, η απέτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια ε, να απαιτούμε δηλαδή δημοσιευμένες πληροφορίες. Έχουμε 6 με 10.000 ε, πράξεις την ημέρα που είναι ηλεκτρονικές. Αν κατάλαβα καλά, η πιλωτική μελέτη που έγινε δείχνει πως ε, μπορούμε να τα λάβουμε αυτά τα, τα δεδομένα. Γιατί να μην είναι συνεχώς προσβάσιμα από την Acer έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να δει τα στοιχεία και να δει μόνος του εάν ε, θεωρούν πως υπάρχει κάποιο μοτίβο ύποπτο. Αυτά τα τρία γενικά μου σχόλια τώρα. Έρχομαι σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον εισηγητή επί των τροπολογιών. Να πω συνολικά πως θεωρώ πως είναι σωστή η κατεύθυνση, το θέμα είναι πως θα το διατυπώσουμε τώρα σωστά. Πρώτα απ' όλα, οι τροπολογίες 2 και 21 αναφέρατε πω πριν υιοθετήσει πράξη τη Κομισιόν πρέπει να συμβουλευτεί του ενδιαφερόμενου. Συμφωνώ. Ποιε είναι οι αρχέ του ενεργειακού τομέα, δεν, δεν καταλαβαίνω τι εννοούμε εδώ πέρα. Τροπολογία 5, ένα γενικό σχόλιο, είναι πολύ καλή η τροπολογία. Χρειαζόμαστε μη ε, Ευρωπαίους, ε, μη ευρωπαϊκές εταιρείε, π.χ. η Gazprom όταν λειτουργεί εντός Ευρώπης να τηρεί τη δική μας νομοθεσία. Ε, αυτό το στηρίζω. Τροπολογίες 6, 8 και 14. Αναρωτιέμαι ποια είναι η προσθέμενη αξία αυτών των τροπολογιών. Στην ίδια πρόταση μιλάμε για ατυχήματα και συντήρηση εγκαταστάσεων και προγραμματισμένη, με συγχωρείτε, συντήρηση. Ε, μα εξορισμού τα ατυχήματα δεν είναι ε, προγραμματισμένα και η προγραμματισμένη συντήρηση είναι ακριβώς προγραμματισμένη. Οπότε οι εταιρείε έχουν ένα πρόγραμμα 6-9 μηνών και ε, όσο νωρίτερα το δημοσιοποιήσουν ε, τόσο μικρότερη πιθανότητα στρέβλωσης της αγοράς. Γιατί αν ξέρουμε πως ε, η εγκατάσταση 1 ε, βγαίνει εκτός τον Ιούνιο, μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας και μπορούμε να προβλέψουμε πως σε μια ανοιχτή αγορά θα παραμείνουν σχετικά σταθερές οι τιμές. Γιατί θα ξέρουμε πως θα υπάρχει μια κάποια έλλειψη. Για... Γι αυτό... Γιατί πάνε αυτά τα δύο μαζί. Και τροπολογία 13 και η τελευταία μου ερώτηση. Ε, πρέπει να το βρω όμως. Α, ναι, τα, τα επιέλατων, τα αντεμήνυμης. Συμφωνούμε, αλλά το όριο αυτό θα οριστεί για να εξαιρέσει από τις απαιτήσει αναφοράς εταιρείε οι οποίες λόγω μεγέθους δεν θα επηρεάσουν τις αγορές. Καλό ακούγεται, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για νομοθεσία. Ή πρέπει λοιπόν να οριστεί πιο συγκεκριμένα ή να βρούμε έναν άλλο τρόπο να πούμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι απίθανο να επηρεάσουν, δηλαδή αν ήμουν εγώ μεγάλη εταιρεία θα έλεγα «Α, εγώ δεν θα επηρεάσω την αγορά». Αλλά έχουμε μια αίσθηση του τι θέλετε να πείτε, αλλά πρέπει να το αναδιατυπώσουμε. Ε, πρόκειται περί νομοθεσίας, ε, δεν είναι λόγια. Σας ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα δικά μου σχόλια. Thank you very much. Ο Dirk Στέρξ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους συναδέλφους. Θέλω να πω ότι μπορώ να τον ακολουθήσω στη γραμμή του τον εισηγητή και είναι και ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το φέρνει αυτό επιτάπητος. Είναι σαφές ότι χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά ε, για να έχουμε μια εύρυθμη, καλώς λειτουργούσα αγορά ενέργειας ε, στην Ευρώπη και όλοι να συμμετέχουν, ε, οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή περίπου όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα και περίπου Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ λίγος ανταγωνισμός στην αγορά. Ένας ε, παίκτης, μία εταιρεία κυριαρχεί και ε, ε, στην προμήθεια φυσικού αερίου και στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στρεβλά που κυριαρχούν στην αγορά και να τα αποκλείουμε όσο γίνεται. Ε, ε, ο εισηγητής στην Επιτροπή Ενέργειας, το είπε και ο κύριος Γκέμπελς, ε, προτείνει κάτι ενδιαφέρον. Να δούμε πώς συνδέεται αυτό με το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων, ETS. Πρέπει να το συνδέσουμε, ναι ή όχι, με ποιο τρόπο. Υπάρχει υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκεί, ή της δικής μας αρκεί να το λέει ο εισηγητής της Επιτροπής Ενέργειας αξίζει να τον υποστηρίξουμε πρέπει να το συζητήσουμε ε, και να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Το κάνει άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει σύνδεση. Ο όρο de minimis είναι κατ' εμέ και απολύτω απαραίτητο. Και το διασυναριακό στοιχείο ενδεχομένω να μπορούσαμε να το προσθέσουμε εδώ, γιατί Νομίζω ότι η αρχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα τις επιμέρους διατυπώσεις, εντάξει. Συμφωνώ και αυτό που είπατε για τις κυρώσεις. Θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Να μην πούμε ότι οι εθνικές κυρώσεις αρκούν. Όχι, να βάλουμε κι εμείς ένα κατόφλι. Τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο. Ε, αλλιώς ε, θα δημιουργήσουμε μια αγορά όπου πρέπει, ο καθένας θα μπορεί να πηγαίνει να επιλέγει ε, πού είναι πιο φτηνά, πού το συμφέρει και θα υπάρχει ένα είδος ε, διαιτησίας. Ως κοινοβούλιο θα πρέπει λοιπόν να πούμε την άποψή μας και να δράσουμε και αν πρέπει να δημιουργηθεί οργανισμός και προσωπικό και πόροι κτλ. Ένα τελευταίο και μετά θα σταματήσω. Ε, στην υποχρέωση κοινοποίηση και ενημέρωση υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται αυτόματα. Αλλά και στο τρίτο ενεργειακό πακέτο έχουμε τέτοιες ρυθμίσει προσοχής στι επικαλύψεις. Στο διπλασιασμό ή και στον τριπλασιασμό να μην χρειάζονται διπλές και τριπλές καταχωρήσεις και κοινοποίησεις όταν κάπου κοινοποιείται κάτι να πηγαίνει παντού όπου πρέπει. Γενικά νομίζω είναι καλή πρόταση και εμείς ως Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τον εισηγητή της Επιτροπής Ενέργειας μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση αυτή και ε, γενικώ συμφωνούμε. Τώρα είναι επιμέρους αυτά διευθετήσεις και αποχρώσεις. Δεν νομίζω υπάρχει κανένα πρόβλημα συνεργασία με τους κοιόδους ηγητές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Uh, ευχαριστώ πολύ. Έχω κι εγώ να πω δύο λόγια. Εδώ και καιρό έχω αποφαθεί γι' αυτό όταν μίλησα για τις διαβουλεύσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντίστοιχη οδηγία. Και νομίζω ότι ό,τι είχα πει τότε έχει καλυφθεί πλέον. υπάρχουν και κάποιες απόπειρες ε, χειραγώγησης και πραγματική χειραγώγηση. Δεν ξέρω αν κάνω εγώ λάθος. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι ή να είπα κάτι λάθος. Εγώ γενικά συμφωνώ ότι η κατεύθυνση που έχει ε, δώσει ο εισηγητής είναι καλή και γενικά είμαι αρκετά ευτυχής. Ρομπέρ, θέλεις να μιλήσεις ξανά εσύ τώρα? Ρομπέρ Γκέμπελς, ναι κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ βεβαίως με τα όσα είπατε και με τον συνάδελφο Στέρξ για αυτό το θέμα της ανάγκης να συμπεριληφθούν ή όχι σε αυτή τη σύσταση ε, οι πολισίες των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, το ETS. Εγώ δεν το έκανα αυτό, γιατί εμείς η, Επιτροπή μας γνωμοδοτεί και μόνο. Και ξέρω ότι ο αρμόδιος εισηγητής στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή το αναφέρει αυτό. Και ε, δικό του θέμα είναι να το συζητήσουν και να εγκρίνουν, να θέλουν ή να μην εγκρίνουν ε, τη συμπερίληψη του ETS. Η χθεσινή συζήτηση έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σκέφτεται και ότι θα ήθελε μάλλον να συμπεριλάβει το ETS στην οδηγία την, την άλλη για την κατάχρηση της αγοράς που χρειάζεται αναδιατύπωση ή μια άλλη για το MIFID. Πάντως αυτή η συζήτηση πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή ως Κοινοβούλιο να ασχοληθούμε ε, για να έχουμε και άποψη. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κάριντς για την πολύ θετική του προσέγγιση. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις. Θα επιθυμούσα να απαντήσω εν συντομία. Νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό να εκτελείται η νομοθεσία ε, με ε, όσο λιγότερη γραφειοκρατία γίνεται. Συναντήθηκα λοιπόν με τον ε, εισηγητή της Καθήλυνα Αρμόδιας Επιτροπής, τον κύριο Χατζημαρκάκη, την ΕΡΓΕΚ που είναι ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστής αυτών των θεμάτων. Πριν δημιουργηθήκαν ο οργανισμός, ε, είχαν κάνει ήδη ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ε, τη ε, διακίνηση της ενέργειας και έχουν αποδείξει ότι όλα αυτά είναι εφικτά. Δηλαδή, τι έδειξαν ότι εάν η αγορά ενέργειας παίξει με τους σωστούς κανόνες στο παιχνίδι, ε, μπορεί να είναι πιο απλοποιημένη η ε, εφαρμογή όλων αυτών με λιγότερο κόστος για τους φορείς και λιγότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Έχει δημιουργήσει και λογισμικό για την υπόθεση αυτή που δείχνει ότι μπορούμε ε, πολύ αποτελεσματικά να εντοπίζουμε όλες τις ανομαλίες στην αγορά. Σας δείχνω τώρα κάποια στοιχεία από εκεί, δεν βλέπετε τίποτα, αλλά ε, κατάφεραν ε, να εντοπίσουν τι έγινε φέτος τον Ιανουάριο, όπου ένας φορέας της αγοράς αγόρασε ηλεκτρική ενέργεια γνωρίζοντας ότι την επομένη ακριβώς ένας μεγάλος παραγωγός θα σταματούσε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή είχε πρώτερη γνώση ως μειόφιλε και το βρήκε αυτό το σύστημα. Και σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Κάρινς, 14 ε, τροπολογία και κάποιον άλλο. τι γίνεται μετά από ατυχήματα ή από συντήρηση. Εγώ είμαι πρόθυμος να δεχτώ διόρθωση της διατύπωσης αυτής, αλλά είναι σημαντικό να υποχρεώσουμε τους μεγάλους παραγωγούς να λέγουν ότι βεβαίως υπήρξαν ε, ατυχήματα ή ότι θα γίνουν επισκευές, γιατί αυτό επηρεάζει και τις τιμές. Σήμερα, αν είναι ένα ίσον ατύχημα, δεν αναφέρεται. Αν γίνει τίποτα τεράστιο σαν τη Φουκοσίμα βεβαίως θα βγει μέσα στον τύπο. Αλλά υπάρχουν ατυχήματα λιγότερο σοβαρά που έχουν επιπτώσει στην παραγωγή ενέργειας και στη μεταφορά ενέργειας. Είτε αυτή είναι ηλεκτρική ενέργεια είτε είναι φυσικό αέριο που δεν κοινοποιούνται αναγκαστικά αλλά που μπορούν να επηρεάσουν, να στρεβλώσουν την αγορά. Εξού και η ανάγκη να ζητούμε πλήρη διαφάνεια και στις ε, ε, εργασίες συντήρησης και σε ενδεχόμενα ατυχήματα. Και είμαι στη διάθεση του αδέλφου Κάρινς για να βελτιώσουμε τη διατύπωση αν δεν του αρέσει ε, η δική μου. Για τον κανόνα de η τροπολογία μου αναφέρεται στο άρθρο 7, όπου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάλλον όχι, να το πω αλλιώς. Προτείνεται ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε κατεξουσιοδότηση πράξης και ε, το ίδιο να ισχύει για τον κανόνα de Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιο είναι το απαραίτητο κατόφλι. Συμφωνώ όμως με τον Dirk Sterks ότι όντως θα χρειαστεί ένα κατόφλι έτσι ελάχιστο έτσι ώστε η πολύ μικρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκείνοι που δεν επηρεάζουν την αγορά λόγω του μεγέθους τους, να ε, προστατεύονται. Ενώ ένας ε, μεγαλέμπορος τύπου Gazprom και τα λοιπά, ε, κολοσσοί τέτοιου τύπου πάντα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την αγορά. Αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας όλων των συναδέλφων για να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλή δουλειά γρήγορα πρέπει να δουλέψουμε γιατί η Επιτροπή Βιομηχανίας έχει ορίσει ήδη χρονοδιάγραμμα. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά είναι αρκετά κοντά. Thank you very much. I'll just read... Ευχαριστώ. Θα διαβάσω τώρα το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μέχρι τις 18 Απριλίου, 3 η ώρα. Δεν γίνεται πιο μετά γιατί πρέπει να κατατεθούν την ίδια μέρα για να έχουμε και τις προθεσμίες της Επιτροπής Βιομηχανίας και επειδή ταξιδεύουν οι συνάδελφοι είναι 3 η ώρα 9 Μαΐου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε επίσης γιατί ψηφίζουν στην ε, αρμόδια επιτροπή 26 Μαΐου και μετά πάει στην ε, δεύτερη ολομέλεια του Ιουνίου. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν πολύς χρόνος και λίγη συνεδρία. Ευχαριστώ τους Γερμανείς.